Colleagues, can I bring the meeting Μήπως μπορούμε να αρχίσουμε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά ψηφοφορίες. Μερικές είναι πολύπλοκες, άλλες ελπίζω όχι. Πριν από αυτά όμως, οι ανακοινώσεις ε, μαζί με τον ορισμό των εισηγητών και συντακτών. Η έκθεση της κυρίας Ράνερ θα εξεταστεί το πρωί και όχι το απόγευμα. Όσοι παρακολουθείτε λοιπόν την έκθεση αυτή να το ξέρετε. Το πρωί και όχι το απόγευμα. Ευχαριστώ την κυρία Ράνερ για την ευελιξία της. Λοιπόν, πάει και αυτό. Ανακοινώσεις. Οι συντονιστές και οι συντονίστριες συναντήθηκαν εχθές το βράδυ και ε, συζήτησαν το θέμα της μαύρης λίστας της Κομισιόν για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τα εμπιστευτικά έγγραφα Δεύτερον, η αποστολή στην Ουάσιγκτον έκανα μια λεπτομερή αναφορά της επίσκεψης και των θεμάτων που συζητήθηκαν εκεί με τα Υπουργεία Μεταφορών και Δικαιοσύνης, βουλευτές και λοιπά. Και οι συντονιστές είπαν να υπάρξει, να προβλεφθεί μια διαδικασία γενικά για τη συνέχεια τέτοιων επισκέψεων έτσι ώστε με τη συνθήκη της Λισαβόνας πια να ξέρουμε τι μας γίνεται. Για την Ουάσιγκτον όμως συγκεκριμένα θα γίνει γραπτή έκθεση αναφορά και θα κυκλοφορήσει, θα μοιραστεί στα μέλη ορισμός εισηγητών και εισιτριών καθώς και συντακτών και συντακτριών. Μία μόνο, ένας μόνο ορισμός. Για έναν κανονισμό που τροποποιεί μια οδηγία για τα στατιστικά στοιχεία ως προς τις μεταφορές αγαθών και προσώπων θαλάσσης. Καμιά ομάδα δεν ήθελε να πληρώσει έναν πόντο για έκθεση και γι' αυτό θα την αναλάβει ο πρόεδρος ή κάποιος αντιπρόεδρος. Έγγραφα που λάβαμε. Έκθεση από για πάλι για τη μεταφορά αγαθών δια θαλάσσης αλλά συστήθηκε να μην υπάρξει καμιά συνέχεια γνωμοδοτήσεις για τις βιώσιμες απαιτήσει για τη διατήρηση των πόρων βιομάζης. Και πάλι, καμία συνέχεια. Τα ίδια και για πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για τη διαχείριση, ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτήων περιοχών. Και πάλι τα ίδια λοιπόν, καμία συνέχεια. Μετά για τις ε, προτάσεις της ΣΤΟΑΣ, ο Κόλ και ο Τρίκα κατέθεσαν τέσσερις συνδυασμένες προτάσεις οριζοντίου χαρακτήρα λέει και αυτές θα εγκριθούν από τους συντονιστές και θα επανυποβληθούν στη ΣΤΟΑ για τελική εξέταση. Οι τέσσερις αυτές προτάσεις αφορούν τη συνεισφορά των λεγόμενων εξύπνων συστημάτων μεταφοράς στην τεχνολογική ανάπτυξη για τη μείωση το, της κατανάλωσης καυσίμων στις θαλάσσιες μεταφορές, ευξημένα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και προκλήσεις στην ε, ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων μεταφορών, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Αυτά ήταν οι τέσσερις προτάσεις της Επίσης συζητήσαμε ένα σχέδιο ψηφίσματος για την εφαρμογή της πρώτης ιδεοδρομικής δέσμης μετά τη συζήτηση της 9ης Μαρτίου. Και οι συντονιστές συμφώνησαν να αναλάβει η Επιτροπή μας ένα ψήφισμα που θα συζητηθεί καταλήλως και θα καταλήξει τον Ιούνιο στην Ολομέλεια η ανακοίνωση μιας κοινή θέσης για δικαιώματα επιβατών θαλασσίων συγκοινωνιών έχουν υποβληθεί τα δύο αυτά θέματα και προβλέπονται στη μήνυ Ολομέλεια και οι δύο εισηγητές θα έχουν την άδεια να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με βάση την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου έτσι ώστε και οι δύο προτάσεις να συζητηθούν μαζί. Μετά έγινε ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης MOVE και προτάθηκε να αναθεωρηθεί η πολιτική της Γενικής Αυτής Διεύθυνσης ώστε να συμφωνεί με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές και μετά τις διαβουλεύσεις η Κομισιόν καθόρισε έξι ομάδες εμπειρογνωμόνων για διάφορες, έξι δηλαδή, πτυχές του θέματος μεθοδολογία, σχεδιασμό, ολοκλήρωση των ε, συστημάτων μεταφοράς, χρήση νέων τεχνολογιών, σχέσεις με τρίτες χώρες ως προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα κλπ. οι ομάδες αυτές εμπειρογνωμόνων θα υποβάλουν τα συμπεράσματά τους στην Κομισιόν και θα καταλήξουν όλα αυτά σε ένα έγγραφο αρχές Μαΐου μεθοδολογικό. 8 9 Τελικά εμείς θα το συζητήσουμε τον Ιούνιο και οι συντονιστές και συντονίστριες της Επιτροπής ΜΕΤΑΦ, τραν δηλαδή, θα τηρούνται ενήμεροι μετά. Αυτά είπαν οι συντονιστές, αφού όρισαν και οι συγητές και συντάκτες και συντάκτριες. Εντάξει, τα δέχεστε όλα αυτά. Σας κατευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και τώρα οι ψηφοφορίες. Πρώτα και καλύτερα παρακαλώ να ελέγξετε αν έχετε φέρει τις κάρτες μαζί σας. Έχουν όλοι και όλες. Εάν τις έχουν παρακαλώ να τις τοποθετήσουν στη σχισμή για να κάνουμε μια, έναν έλεγχο. Βλέπω τον κύριο Στύρκ να παλεύει εκεί. Λοιπόν, Έλεγχος άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Μαγδαληνή ε, στείλε κάποιον να στη φέρει. Ή κάποιον. Έληξε η δοκιμαστική ψηφοφορία. Έληξε. Εντάξει ήτανε. Τα κοιτάξατε. Ο κύριος Στέρξ είναι πάντοτε ο κύριος Στέρξ και κατά την ψηφοφορία μάλιστα. Δύο βουλευτές δεν έχουν τις κάρτες τους. Μήπως και κανείς άλλος δεν την έχει για να τους λάβουμε υπόψη κατά τις ψηφορίες. Υπάρχει η κυρία Αλβάρες και ο κύριος Κράμερ. Λοιπόν, μάλιστα. Αρχίζει το rock τώρα. Λοιπόν, πρώτον το σχέδιο έκθεσης για ό,τι ισχύει για τα πλοία που αποπλέουν και καταπλέουν σε κοινοτικού λιμένες. Έκθεση του κυρίου Στέρξ. Ένα. Προπολογία 44 του κυρίου Μαρινέσκου. Υπέρ. Κατά. Ποιες. Απαρρίπτεται. Δεν χρειάζεται έλεγχος. 14 του εισηγητή υπέρ τα και εγκρίνεται. 45 δεν θα αναφέρω τα ονόματα των συντακτών, με συγχωρείτε για να είναι πιο γρήγορα. Λοιπόν, μετά θα γίνουν πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Λοιπόν, 45 Μαρινέσκου, ορίστε θα τα λέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απαρρίπτεται. 46 Μαρινέσκου, υπέρ. Κατά. Χες. Απορρίπτεται. 47 Μαρινέσκου, υπέρ. Κατά εποχές παρύπτεται. 15 του εισηγητή με προφορική τροποποίηση του ιδίου. Την έχετε εδώ μπροστά σας, την τροποποίηση υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται 48, έχει αποσυρθεί. 16 του εισηγητή υπέρ, τα Ποιες γκρίνεται 17 εισηγητή. Ε, υπερκατά. Ποιες. Όχι, επαλήθευση. Επαλήθευση για τη 17 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία η κυρία Αλβάρες και ο κύριος Κράμερ θα μας πούν προφορικά. Έληξε η ψηφοφορία. Υπέρ 16 κατά. Εγκρίνατε λοιπόν. Ήσασταν κατά. Α, 21 προς 17 λοιπόν. Εκείνος που δεν έχουν τις κάρτες τους. Τον παρακάτω. 49, μόνο την τελευταία πρόταση, γιατί η 17 έχει διεγκριθεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 50 κατέπεσε. 18 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 και 53 έχουν αποσυρθεί. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Στέρξ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 20 έχει αποσυρθεί. 54 στέρξ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 για το άρθρο 7α νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη 57. 57. Τεγράδες Πασκουάλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 το εισηγητή υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι είναι κρίθη αλλά για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά και την 24 ελέγχουμε ψήψαν όλοι πέρας 22 υπέρ 14 κατά Εγκρίνεται λοιπόν. 25 Πενήντα 58 στέξ με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Και με την αδειά σας θα ψηφίσουμε την 59, 61, 62, 63, 11, 61 μαζί με την 58. Γιατί όλες το ίδιο είναι. Μπορούμε να συμφωνήσουμε on block αυτές τις πιστοπολογίες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. 26 εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 μπάσετ υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 60 παρακαλώ ελέγχουμε ηλεκτρονικά ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας η κυρία Αλπέρης είναι υπέρ Μάικλ υπέρ 19 υπέρ λοιπόν 18 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Fall, so we know... 28 καταπίπτει. 1 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 πίπτη. συμβεστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 3 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 καταπίπτει εκτός από εκείνο που λέει ε, αστυνομία Συνόλου και Ευρωπόλ. Θα ψηφίσουμε αυτό σαν προσθήκη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα του εισηγητή, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 πρώτο τμήμα. Έχει καταπέσει για την με του 51. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερη πρόταση δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 32 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 22 υπέρ 14 κατά, ναι, είναι κρίθη. 7 έχει χρήση 34 στέρξ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Την 5 και 8 έχουν καλυφθεί. Η 9 έχει εγκριθεί αυτόματα γιατί εγκρίναμε τη 17. 36. Έχει καταπέσει. 38 έχει αποσύρθει. Δεν σας είπα ότι περιπλέκονται τα πράγματα. 39. Τεγράτες Πασχουάλ, Βλάσκο κλπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Βαντάλεν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ελέγξουμε. Την 10 του εισηγητή. Άρχεται ψηφοφορία. Τώρα έχετε την κάρτα σας κυρία Αλβάρες; Ωραία, πέρασε ψηφοφορίες. 19 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 40 έχει αποσυρθεί. Την 11 έχει καλυφθεί ήδη. 13. 13. Του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και 42 φαντάλλων. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται επίση. Τελική ψηφοφορία για την νομοθετική πρόταση ως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Και την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχιε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Ανεκρίθη επίσης. Συγχαρητήρια για τη στέρξη. And Mr. Kramer in favour. Thank you, Michael. Next Επόμενο. Ψηφοφορία. Για, τη μεταφορά εξοπλισμού υπο... για υλικό υποπίεση. On block, συμφωνείτε, να ψηφίσουμε όλες μαζί. Αν όχι θα πρέπει να τις μία-μία-μία. On Σήμερα Συμπεριλαμβανομένες και τις προφορικές τροπολογίες για 43. Ωραία. Όλα on block. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Εγκρίνονται. Ναι. Νομοθετική πρόταση. Α, όχι. Έχουμε και μια προφορική τροπολογία υπαριθμών 6 που πρέπει να εξετάσουμε ξεχωριστά. Μια νέα προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, απαχές Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 35 mm. υπέρ, Καμία ψήφος κατά. Δύο αποχές. Νομοθετικό ψήφισμα. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34-02. Εγκρίνεται λοιπόν. And στην επόμενη έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τους στρατηγικούς στόχους και συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018. Η εισηγητής ο κύριος Βαντάλεν. Ξεκινάμε με την παράγραφο 1, τροπολογία 11 του κυρίου Τούσα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 για λασέντερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 τούσας, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 της κυρίας Τσικάου υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. 14 της κυρίας Τσικάου. Άρχεται η ψηφοφορία. Μάικολ, να μας πεις τι θα ψηφίσεις. Πέραση της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. 15 Μπέσετ υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, urges the commission, flags of convenience, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε το πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε και την ψήφα του κυρίου Κράμερ. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. End to look μέχρι register. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Μία ψήφος υπέρ από τον κύριο Κράμερ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας στις ψηφοφορίες. 13 υπέρ, 26 κατά απορρίπτεται. 17 του κυρίου Τούσα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τοπολογία α, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 του σας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 Βλάστο Ρίκετ κατά τμήματα πρώτο τμήμα από Considers That μέχρι Applicable Legislation υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα Ισχύει notes that μέχρι του restrictive υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 για λασέντερ υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. 23 του κυρίου Κουμουτσάκου κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, το σύνολο του κειμένου χωρίς το end extended, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν, το end extended, υπέρ, κατά, αποχές. Να κάνουμε έναν έλεγχο με την προσθήκη των δύο αυτών λέξεων. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορία. 25 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. 24 μπέσετ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Φλέκενστάιν. Έχω και μια προφορική τροπολογία του εισηγητή εδώ. Κύριε Βαντάλεν. Mm. Κύριε Πρόεδρε. Τώρα το κείμενο λέει, μιλάει για Αύγουστο 2010. Νομίζω πρέπει να πούμε απλώς 2010 χωρίς μήνα. Και άνευ μηνός. Εκτός μικροφώνου είναι ο Πρόεδρος. Α, με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. 26. Ο κύριος Φλέκενστάιν, προφορική τροπολογία από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κύριε Φλέκενστάιν. Ναι, αντικαθιστούμε το safeguarding με το promoting και προσθέτουμε και να διασφαλίσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Αν όχι, ψηφίζουμε μαζί με την τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 του κυρίου Φλέκενστάιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι, βλέπω ότι βαριέστε να σκώσετε τα χέρια σας. 28 Φλέκενστάιν. Κατά τμήματα, πρώτο τμήμα μέχρι το short shipping υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, calls on the community υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, 29 του σας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 34 του κυρίου Κουμουτσάκου. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι το Maritime Colleges υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, at the same time μέχρι with fatigue, υπέρ, κατά, αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της 34, άρχεται η ψηφοφορία. Κύριε Κράμερ, είστε υπέρ. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. Η 33 καταπίπτει. Συμβιβαστική τροπολογία C. Έχουμε μια συμβιβαστική τροπολογία με κατατμήματα ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία, πρώτο τμήμα μέχρι το Necessary Assisted by Ensem. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με τη φράση αυτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάει η συμβαστική τροπολογία λοιπόν στο σύνολό τη. 36 Μαρινέσκου. Περ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έναν έλεγχο. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε τη 36. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο Μάικολ είναι κατά. Πέραση της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 37 Μαρινέσκου υπέρ, κατά, Αποχές συγκρίνεται. 38 καταπίπτει. 41. Ο κύριος Φλέκενστάιν και πάλι μια προφορική τροπολογία από τους ελστές και δημοκράτες. Ναι, αντικαθιστούμε το review με το extend. Αυτό. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές να κάνουμε μια επαλήθευση. Νομίζω ότι απορρίπτεται να ψηφίσουμε τη 41 με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Όντως απορρίπτεται 15 υπέρ 24 κατά. Δεύτερο τμήμα τη 43. Το πρώτο τμήμα καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία C. Το δεύτερο τμήμα με το particularly important issue κλπ. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44. Βλάστορικέ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 45 λοιπόν καταπίπτει, 46 σας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 και υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ. Ποιος θα τα πει. Ο κύριος Κομουτσάκος. Στην ε, προφορική μας τροπολογία υιοθετούμε μια λιγότερο δεσμευτική γλώσσα από ό,τι είχε αρχικώς προταθεί ε, και ενώ διατηρούμε ακριβώς το ίδιο πνεύμα της προταθής αστροπολογίας απλώς η φρασιολογία με την ε, προσθήκη «in this respect ε, will be of particular interest» είναι μεγαλύτερης ευελιξίας και νομίζω ότι μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ ενστάσεις για την προφορική τροπολογία. Αν όχι, την ψηφίζουμε μαζί με την 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυτή είναι η ίδια. Είναι συμβατή με την 52. Θέλετε να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 Κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, το σύνολο του κειμένου χωρί τη φράση πριν από το τέλος του 2010, το δεύτερο τμήμα θα περιλαμβάνει και αυτή τη φράση. Το πρώτο τμήμα λοιπόν χωρί αυτή τη φράση, υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα, με τη φράση, υπέρ. Καταπίπτει ούτως ή άλλως. Καταπίπτει, συμφωνούμε. Δεν ψηφίζουμε τίποτα άλλο. 55. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το σύνολο του κειμένου χωρίς τη φράση αυτή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έναν έλεγχο παρακαλώ. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα της 55. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. So we don't do the second part then. Second part. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 56 κούν υπέρ. Κατά. Αποχές εκρίνεται. 57 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 του κυρίου Κούν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα considers that all με external costs υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα believes that μέχρι το innovation υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κύριε Γκρός. Κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουμε πρώτα τη συμβιβαστική τροπολογία D και μετά να αποσύρουμε τις 63 και τις 64, εάν περάσει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτή τη ψηφοφορία. Ωραία. Θα ψηφίσουμε πρώτα τη συμβιβαστική τροπολογία D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. η συμβαστική τροπολογία ήταν, έπρεπε να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα, συγγνώμη δικό μου λάθος, έπρεπε να ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου χωρίς τη φράση και να αναλύσουν τα έξοδα λιμένους. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 1423. Δεύτερο τμήμα με τη φράση αυτή. Θα ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικός. Δεν... Συμβαστική... Α, δεν έχει πλέον νόημα. Ε, δεν υπάρχει συμβαστική τροπολογία D, 63 και 64, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. Ψηφίζουμε τώρα την 65 του κυρίου Κουμουτσάκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κύριε Στέρξ. Τι έγινε με τις 63-64, απορρίφθησαν. Παράγραφος 16 έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από το ΕΛΚ για την παράγραφο 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67. Κύριος Σκούν. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70. Προφορική τροπολογία από το ΕΛΚ. Κύριε Κουμουτσάκο, παρακαλώ.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 κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 της κυρίας Τσικάου υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έναν έλεγχο. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά προτιμώ να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 76. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 15 με τον Μάικολ, 23 κατά. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία Ή. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 είναι η επόμενη, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα μέχρι το Transport System, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη, δεύτερο τμήμα, έχει νόημα, έχει, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 ως προσθήκη συμβιβαστική τροπολογία ή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 της κυρίας Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 99 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στα εκτιμώντα 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, να κάνουμε έναν έλεγχο για την 4, βλάστορη και υπέρ, άρχεται ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας τη ψηφοφορία. 19 υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται, επομένως καταπίπτει 5, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έναν έλεγχο για την 9 παρακαλώ επαλήθευση της 9 βλάστορη και άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Mm. Πέρασε της ψηφοφορίας. Mm. 19 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 10 της κυρίας Τσικάου, υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Ζητά, ζητείτε έλεγχος για τη 10, Τσικάου, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. 14 υπέρ 22 κατά πράγματι απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ευχαριστώ. Πέρασε τη ψηφοφορία. Υπέρ ο κύριο Κράμερ. 34 υπέρ, 1 σκατά και 3 αποχέ. Χαρητήρια λοιπόν στον κύριο Βαντάλεν. Πέρασε η εκθεσή σας. Τώρα, η γνωμοδότηση για τη στρατηγική για τη Βαλτική. Έκθεση, ε, γνωμοδότηση Κουν, Βέρνερ Κουν μάλιστα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά τη χθεσινή συζήτηση, από πλευρά ΣΕΝΚΑ θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι Τροπολογίες 6, 15 και 16 μπορούμε να τις δεχτούμε. Να έχετε μαζί δηλαδή στη λίστα κάτι ψηφοφορίας. So that's for the EP. Α, για το ΕΛΚ αυτά. Να αλλάξετε τον κατάλογο ψηφοφορίας σας. Λοιπόν, Αρχίζουμε με την παράγραφο 2 τροπολογία 1 του κ. Μπαλτσέιτης υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 ζήλε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι εκεί που λέει τέν τάφ 21 υπέρ κατά αποχές απαρρίπτεται δεύτερο τμήμα έχει νόημα εντάξει δεύτερο τμήμα υπέρ τα χες εγκρίνεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 next yeah 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 ζήλε υπέρ τα χες εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 10 Άουκεν υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για τη 10 ηλεκτρονικός. Άρχισε η ψηφοφορία ήδη. Ψήφισαν όλοι και όλες. Έληξε. 21 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 11 Φλέκενστάιν με προφορική τροποποίηση του συγκριτού κυρίου Κούν. Θέλουμε να αντικατασταθεί εκεί που λέει shipping links must be promoted in order to ensure efficient use of the sea. Να αντικατασταθεί η προηγούμενη διαβτύπωση από αυτήν. Μάλιστα, με αυτή την τροποποίηση λοιπόν υπέρ της 11 κατά ποιες γκρίνεται 12 υπέρ τα ποιες γκρίνεται 13 υπέρ κατά ποιες γκρίνεται 14 υπέρ κατά εποχές επαλήθευση για τη 14 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι και όλες έληξε 14 υπέρ 23 ε, κατά απορρίπτεται 15 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 16 υπέρα. Πώς, πώς. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, επετάξαν πολλές καλές συμβαστικές λύσεις και η συζήτηση στην Επιτροπή χθες κατέδειξε ότι η ε, ανάπτυξη των ε, ε, διαδρόμων για ποδήλατα θα πρέπει να βελτιωθεί και γι' αυτό θα ήθελα για τους στόχους αυτούς να υποστηρίξουμε τη σχηνική τροπολογία και γι' αυτό σας παρακαλώ να υποστηρίξετε Okay, Amendment 16. Those in favor. Those against. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Επαλήθευση για, τις δεκα, για τη 19 ζήλε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εάν ψήφισαν όλοι και όλες έληξε η ψηφοφορία. 20 υπέρ 18 κατά εγκουρίνεται. Τελική ψηφοφορία, συνολική. Ηλεκτρονικά, άρχεται. Ο κύριος Κράμερ είπε υπέρ. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Έληξε η ψηφοφορία 36 υπέρ, μία ψήφος ε, κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Κούν μου. Και τώρα συνάδελφοι έληξαν οι ψηφοφορίες. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Επόμενο θέμα είναι, είναι λέγω, το Ευρωπαϊκό Συνδρομικό Δίκτυο για Ανταγωνιστικές Εμπορευματικές Μεταφορές. του κυρίου Μαρινέσκου. Τσακ τσακ. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Όπως πάντοτε όσοι θέλουν να φύγουν να διαλυθούν ηρέμως. όσοι δεν θέλουν να μείνουν να μείνουν επίσης ηρέμως. για να ακούσουν τον εισηγητή. Χωρίστε κύριε Μαρινέκου. Ευχαριστώ κύριε Όπως μετά από τις διαβουλεύσεις που έκανα κατέθεσα τις τροπολογίες που θεωρούσα απαραίτητες προς τον κανονισμό αυτόν. Είχα μία πρώτη συνάντηση με την Ισπανική Προεδρία και καταφέραμε να εξετάσουμε ολόκληρη την έκθεση μαζί. Ολόκληρη, όχι κατά τμήματα. Θα ήθελα να σας αναφέρω που πρέπει να συζητηθούν ορισμένα σημεία περαιτέρω. Γενικά θα συμφωνήσουμε μου φαίνεται για πολλά σημεία του κειμένου, αλλά υπάρχουν και τρία όπου θα χρειαστεί περαιτέρω διαπραγμάτευση. Πρώτον, το One Stop Shop, δηλαδή ο τόπος όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσει για να περνάει η ενιαία σιδηροδρομική γραμμή διαμεθοριακά. Σας παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος να μην κάνετε πηγαδάκια εδώ μέσα, είναι αγενές αφού ο εισηγητής προσπαθεί να μας εκφράσει την έκθεσή του. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε και να συνεννοηθείτε, αλλά υπάρχουν τεράστιοι διάδρομοι γι' αυτό και παρακαλώ να σέβεστε τον εισηγητή που κάνει την προσπάθειά του. Ορίστε κύριε Μαρινεύκο. Λοιπόν, όπως έλεγα, ένα από τα κύρια φιλεγόμενα σημεία είναι το One Stop Shop. Εμείς διαφέρουμε από την, με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εμείς δηλαδή θεωρούμε ότι, ότι και όταν λέω εμείς εννοώ και εμένα και τους σκιώδεις, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το One Stop Shop πρέπει να αποφασίζει, να κρίνει τα αιτήματα. Ενώ το Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό το One Stop Shop πρέπει μόνο να δέχεται αιτήματα και να είναι ένα κέντρο πληροφόρησης. Και μετά να αποφασίζουν οι διευθυντές των σιδηροδρομικών εταιριών των χωρών και εκείνοι να αποφασίζουν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το κύριο θέμα της έκθεσης και η προστιθέμενή της αξία. Γι' αυτό θέλουμε να αλλάξει αυτό το σημείο. Δεύτερο αμφιλεγόμενο θέμα. Οι λεγόμενοι authorized applicants, νενομισμένοι αιτητές. Εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να ζητήσει μια διαδρομή ενώ το Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό θα ισχύει μόνο για ιστορικές και γνωστές σιδηροδρομικές εταιρείες. Να δούμε τι συμβιβασμός μπορεί να πετευχθεί εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε στη θέση μας γιατί εμείς δουλεύουμε σε ανοιχτή αγορά και για τις μεταφορές. Μην το ξεχνάμε. Κάτε με, ο περιορισμός της έγκρισης δρομολογίων μόνο για προεγνωσμένες και ιστορικές εταιρείες στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και την αγορά. Τρίτο αμφιλεγόμενο σημείο, οι προτεραιότητες σε περίπτωση των συγκοινωνιών. Συμφωνήσαμε ότι το κύριο κριτήριο για την επίλυση τέτοιων συμβάντων πρέπει να είναι ο ελάχιστος χρόνος επανάληψης των διαδρομών και από εκεί και πέρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να καθοριστούν ορισμένες προτεραιότητες. Κάποιοι όροι, ας πούμε, αν είναι επιβατικό το τρένο που έχει σταματήσει την κυκλοφορία του για 3-4 ώρες, τότε το επιβατικό αυτό τρένο να έχει προτεραιότητα στην επανάληψη. Ενώ το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι χρειάζονται τέτοιοι κανόνες προτεραιότητας. Και υπάρχει και άλλο τέταρτο εμφυλεγόμενο σημείο, πιο γενικό όμως, γιατί αφορά ολόκληρο το έγγραφο, ολόκληρο, και είναι ο καθορισμός μίας διαχειριστικής επιτροπής από εκπροσώπους χωρών μελών που θα το καθορίζουν οι διευθυντές των συντηροδρομικών επιχειρήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι επιτροπές πρέπει να έχουν ορισμένες προκαθορισμένες ευθύνες. Γιατί αλλιώς όλα θα αποφασίζονται μόνο από τις σιδηροδρομικές εταιρείες ή από τις διαχειριστικές αυτές επιτροπές. στο Συμβούλιο συμφωνεί να δημιουργηθούν αυτά τα σώματα, αυτές οι επιτροπές, αλλά θέλει οι αποφάσεις να λαμβάνονται μόνο από τους διευθυντάς. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβασμό τελικά βέβαια. Αυτά είναι τα κύρια τέσσερα αμφιλεγόμενα σημεία της εκθεσής μου. Νομίζω ότι στη δεύτερη μας συνάντηση θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε όλα αυτά γιατί όπως σας είπα κατά την πρώτη συνάντηση με το Συμβούλιο εξετάσαμε τουλάχιστον τη μισή έκθεση και τώρα θα εξετάσουμε το δεύτερο μισό. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου για τους σοσιαλιστές ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής, ο κύριος Μαρινέσκου, παρακολουθεί το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό πλέον και στη διάρκεια της προηγούμενης Προεδρίας και στην τρέχουσα και ε, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο, στο οποίο πρέπει να αποδεικνύεται η όβιος υπομονή. Και λέω υπομονή διότι η Σουηδική Προεδρία, αν θέλετε, αντιμετώπισε το θέμα εκ του μακρόθεν και τώρα υπάρχει λίγος μεγαλύτερος ενθουσιασμός με την Ισπανική Προεδρία που δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει το θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να ε, ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο στασιμότητας. Τι νέα ποιότητα λοιπόν θα έχουμε με αυτούς τους σιδηροδρομικούς ε, διαδρόμους. Πρόθεσή μας είναι να γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ε, ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. Η πρόθεση όμως του Συμβουλίου είναι να γίνουν μεν πάρα πολλέ κινήσεις, αλλά μόνο για τους τύπους που και στη συνέχεια να έχουμε μια κατάσταση απαράλλακτη με τη σημερινή. Ο κύριος Μαρινέσκου παρουσιάζει ένα πακέτο προτάσεων για θέματα τα οποία εξακολουθούν να είναι υποσυζήτηση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσον έχουμε τις δυνατότητες να ζητήσουμε ε, σωστό καταμερισμό αυτών των εμπορευματικών ε, διαδρόμων. Και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να στοχεύσουμε. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το πακέτο, διότι δίνει προτεραιότητα στις μεταφορές, στην κίνηση ε, και μάλιστα με πιο αποτελεσματικό τρόπο για τους επιβάτες και όχι μόνο για τα εμπορεύματα. Συμφωνώ και με τα όσα λέει ο ε, για, την, ε, για το One Stop Shop θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε και μια ευρύτερη μορφή του One Stop Shop. Η ομάδα μου συμφωνεί και με τον εισηγητή για το θέμα των αρμοδιοτήτων ε, του διευθυντή των υποδομών, του διαχειριστή των υποδομών. Δεν είμαστε εμείς ε, αυτοί οι οποίοι θα ε, δώσουμε δυνατότητα απόφασης στον διευθυντή. Εμείς, όπως είπα, θέλουμε να προσδώσουμε νέα ποιότητα στον τομέα αυτό. Σε γενικές γραμμές, ε, νομίζω λοιπόν ότι οι απόψεις μας ε, συμπίπτουν απόψεις δηλαδή μεταξύ της ομάδας μας και του εισηγητή. Οι προτεραιότητες μας είναι κοινέ. Και ο εταίρος μας και ο αντίπαλός μας ταυτόχρονα είναι το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε κοινό έδαφο συνεννόησης ε, τις, για τις προτεραιότητέ μας με το Συμβούλιο. Θα προσπαθήσουμε όμως να κάνουμε κάποια βήματα υπέρ ε, συμβιβασμού και φαντάζομαι ότι εμείς ως κοιόδης εισηγητή και ο εισηγητή θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ίδια άγουσα. Για τους φιλελευθέρου τώρα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Μαρινέσκου πολύ σωστά επικεντρώθηκε στα θεμελιώδη προβλήματα που έχουμε με τη θέση του Συμβουλίου. Η μία και μόνη θηρίδα, οι προτεραιότητε σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας ε, και ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι επιπλέον. Η διαφορά που έχουμε οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο είναι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου κάτι το οποίο το Συμβούλιο δεν δέχεται. Η πολιτική μου ομάδα θεωρεί ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρομικών διαδρομών, ε, εμπορευματικών διαδρόμων και εδώ θα ήθελα να σταθώ σε μία παράγραφο η οποία προκάλεσε κάποιες συζητήσεις ε, και μάλιστα τις θέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Το ε, κείμενο που μιλάει για τον ορισμό των νέων διαδρομών που κάνει το Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι μέχρι τούδε όταν ε, μιλούσα για το θέμα αυτό σε διάφορες επιτροπές ήμουνα πολύ προσεκτική αλλά μετά από τις διάφορες συνεδριάσεις που έκανα και τις πληροφορίες που έλαβα ακόμα και γραπτός ε, πρέπει να πω ότι υπάρχει απόλυτη έλλειψη διαφάνειας από πλευρά Συμβουλίου στο θέμα αυτό, διότι τους έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να μας δώσουν τα επιχειρήματα ε, για τους λόγους για τους οποίους περιλαμβάνουν αυτούς τους διαδρόμους στο παράρτημα 1 ποιες είναι οι αναλύσεις που διαθέτουν, αν διαθέτουν οικονομικές, κοινωνικές αναλύσεις, ε, ποια είναι τα σημεία στα οποία θέλουν να σταθούν και γιατί περιλαμβάνουν κάποιους διαδρόμους και κάποιους άλλους όχι. Και αν υπάρχει κάποιος μεικτός χαρακτήρας θα πρέπει να μας διευκρινίσουν γιατί συμπεριλαμβάνονται αυτοί οι νέοι διάδρομοι, γιατί πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση πάντα υπό το πνεύμα της ε, προσθήκης ε, και επαναλαμβάνω ότι πρέπει όλοι οι ευρωβουλευτές να έχουμε πληροφορίες για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε και το σχετικό θέμα. Πρέπει να πω ότι μέχρι σήμερα δεν μας έχει δοθεί ουδέμια πληροφορία και το μόνο λογικό επιχείρημα ήταν αυτό είναι αυτό το οποίο υπερασπίζεται κάθε χώρα. Στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε με το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε και επειδή και στο κείμενό της περιλαμβάνονται στα κριτήρια βάσει των οποίων θα εγκρίνονται νέοι διάδρομοι, η Επιτροπή μας είπε ότι οι διάδρομοι που περιλαμβάνονται σε αυτό το παράρτημα, κατά την άποψή τους, καλύπτουν αυτά τα κριτήρια. Εμείς όμως ως Ευρωβουλευτές, υπεύθυνοι για το θέμα αυτό, δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια των κρατών μελών και του Συμβουλίου για να ορίσουν αυτό το πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Ο κύριος Μαρινέσκου ζήτησε εννέα ε, θέματα γραπτός ε, τα οποία απασχολούν εμάς ευρωβουλευτές και δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Στην τελευταία συνάντηση ρωτήσαμε προφορικός και ζητήσαμε να μας δώσουν ε, πληροφορίες και πάλι δεν πήραμε καμία απάντηση. Και εγώ θα ήθελα να σας πω σήμερα ότι οι φιλελεύθεροι έκαναν μια τεράστια προσπάθεια για να συμπεριλάβουν προτάσεις στο κείμενο αυτό. Και για άλλη μια φορά ζητάμε το Συμβούλιο τουλάχιστον να μας ενημερώσει. Ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής. Γιατί θεωρούν ότι με τα κριτήρια αυτά, με αυτούς τους διαδρόμους θα δημιουργήσουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Τι χαρακτήρα έχουν αυτοί οι διάδρομοι τι σχέσεις θα έχουν με τα ε, σχέδια τα οποία είναι εξελίξη και ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Αυτά όλα θα ήθελα να διευκρινιστούν σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Η προθυμία των φιλελευθέρων ε, είναι προφανές ε, με όλες τις προτάσεις που κάναμε στο κείμενο το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο, αλλά θα ήθελα σήμερα επισήμως να ζητήσω για άλλη μια φορά το Συμβούλιο να μας αποστείλει τουλάχιστον τα κριτήρια βάσει των οποίων συμπεριλήφθησαν αυτοί οι νέοι διάδρομοι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριος Κράμερ από τους πράσινους. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου. Είχαμε μια σειρά συναντήσεων και πέρσι και φέτος και Χαίρομαι που δεν έχουμε πια την πίεση χρόνου που είχαμε και μπορούσαμε να το συζητήσουμε αναλυτικά. Εγώ θα ήθελα να μεθεθώ σε ένα θέμα που ήδη εφήγει. Όταν κάπου γίνει ένα δυστύχημα ή μια διακοπή τέλο πάντων τη ε, διαδρομή, εγώ είμαι υπέρ τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Να μην υπάρχει προτεραιότητα για κανέναν. Παραδείγματο χάρη, έχουμε μια οδηγία για του οδηγού των ε, για τους μηχανοδηγούς. Και αν μετά από ένα τέταρτο ή μισή ώρα λίγη ο χρόνος μέσα στον οποίο επιτρέπεται να οδηγήσει ο μηχανοδηγός αυτός, δεν παίζει κανένα ρόλο τι ε, ε, σειρμό οδηγεί εκεί. Ε, εμπορευματικό, ταξιδιωτών κλπ. Θα πρέπει αυτό το τρένο όμως να περάσει το γλυγορότερο δυνατόν στην, ε, στην πρόθεση πρώτο. Αυτό είναι το κριτήριο. Ναι. Δεύτερον, δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών κρατικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επιχειρήσεων. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την, ε, και να ενδυναμώσουμε την εσωτερική αγορά. Θέλω να είμαστε ε, δίκαιοι. Εμείς είμαστε υπέρ των συνδρομών, όχι υπέρ κάποιες συγκεκριμένες συνδρομικής επιχείρησης. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, Μόνο τα κρατικές επιχειρήσεις μπορούν να εισπράξουν κρατικές επιδοτήσεις του φορολογούμενου. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να πληρώσουν από τις τους. Άμα το κάνουμε αυτό έτσι, ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Δεν είναι ποτέ θεμητός και δίκαιος κατά αυτόν τον τρόπο. Επίσης μου φαίνεται προβληματικό το θέμα των ε, ιδιαίτερα σημαντικών ε, διαδρομών. Εγώ ξέρω μόνο μία. Ε, μεταφορές μεταξύ Ρώμης και Νάπολης τη νύχτα. Αυτό ισχύει μόνο για τη νύχτα. Μόνο τη νύχτα μπορούν να ε, κυκλοφορούν εκεί οι σειρμοί που μεταφέρουν αγαθά και όχι την ημέρα. Κατά τα άλλα υπάρχουν πολλές καταχρήσεις, το είπα. Εγώ είχα επεκρίνει μια κρατική επιχείρηση που είχε δηλώσει 20-30 διαδρομές χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία. Τις είχε δηλώσει και καταγράψει μόνο για να μην δώσει ευκαιρία στους αγωνιστές να τις χρησιμοποιήσουν. Η καταγραφή ήταν ατελής. Πόσο πιο φθηνά μπορώ να αποτρέψω τον αγωνιστή μου να μπει στο δίκτυο. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει ένα κόστος για την κράτηση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα οικονομικό αντίκτυπος αν ε, κανένας δεσμεύει ε, ε, διαδρομές και σλότ. χωρί να τα χρησιμοποιεί. Όσον αφορά τον ρυθμό των διαδρόμων, δεν κατάλαβα γιατί έχετε διαφορετικό αποτέλεσμα. Όταν κάνουμε μια ανάλυση γιατί από τους έξι διαδρόμους αυτούς δεν έγινε τίποτα, πώς μπορεί να μου είπε κανένας ότι δεν μπορέσαμε να τους πραγματοποιήσουμε τα προηγούμενα χρόνια και τώρα ε, χρειαζόμαστε όμως ε, εννιά. τι σας πω, εγώ δάσκαλος είμαι, αν μας μου έλεγε τέτοιο πράγμα, θα είχε αποτύχει αμέσω. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε έναν από τους διαδρόμους αυτούς, ούτε τον Α που είναι ο πιο σημαντικός στην Ευρώπη. Λοιπόν, ας κάνουμε άλλη συζήτηση για νέους διαδρόμους μετά που θα έχουμε συγκεντρώσει προσοχή μας αυτού που έχουμε ήδη αποφασίσει. Περίεργο μου φαίνεται επίση ότι πρόκειται για διαδρόμου. Ένα έχει καθαριστεί όμω. Στοκχόλμη και ε, Τζένοβα. Στοκχόλμη, Κοπενχάγη, Αμβούργο, Ίντσπρουκ και διαμέσω τίποτα. Γιατί να έχει ε, ε, αποφασιστεί κάτω αυτού κάτι τέτοιο αυτό είναι μόνο για, τον, <clears throat> για την γέφυρα στη Φέμανα πάνω στη Γερμανία που έχει αποφαστεί χωρίς να αρχίσει να χτιστεί. Δεν ξέρουμε καν πότε θα χτιστεί, αν θα είναι τούνελα, αν θα είναι ε, γέφυρα. Καθορίζεται αυτό, αλλά παραβλέπουμε το πιο σύνομο δρόμο θεωρών Ρόστοκ, Κοπενχάγη. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Μετά, τα one-stop shop. Γιατί θέλουμε μία ευρωπαϊκή οργάνωση που καθορίζει τα πάντα. Γιατί τι θα κάνει αυτή. Θα ρωτήσει εθνικές επιχειρήσεις, έχετε κάποια σλότ ε, ε, ελεύθερα. Εγώ αυτό φανταζόμουν σε ένα λεγόμενο πραγματικό one-stop shop, ότι εγώ ας πούμε ε, είμαι πελάτης και θέλω να μεταφερθώ από το Rotterdam στην Τζένοβα. Ρωτάω κάποια συγκεκριμένα υπηρεσία και μου λέει εκείνη, η οποία έχει σε επαφή με όλε τι διάφορε χώρε. αν είναι δυνατόν να εγκριθεί. Εάν εγκριθεί, εγκρίνεται. Αν δεν εγκρίνεται, μπορεί να υπάρχει κάποια υπηρεσία διατησίας ευρωπαϊκή που θα λέει τι έγινε, ποιος προτιμήθηκε κλπ. Θέλω να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Για τον πελάτη θα πρέπει να είναι σαφές γιατί αυτή η υπηρεσία, η ευρωπαϊκή αυτή η υπηρεσία θα γνωρίζει όλα τα επιχειρήματα, όλα τα κόλπα, πώς μπορεί να αποφύγει κανένας τους ανταγωνιστές του. Πάνω σε αυτό θα μπορούσα να συμφωνήσω με ένα συμβιβασμό νομίζω. Όχι μια τεράστια γραφειοκρατία, δηλαδή καινούρια, αλλά κάποιον συνομιλητή για τους πελάτες, για την Ευρώπη. Γιατί κάνουμε εδώ ευρωπαϊκή και όχι εθνικιστική πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Κούν. Oh, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ταιριάζει αυτό. Γιατί καταρχήν θα ήθελα να διορθώσω τον κύριο Κράμα στη Γερμανία οι κρατικές επιχειρήσεις δεν παίρνουν για, την, ε, <clears throat> τη λειτουργία τους επιδοτήσεις, μόνο για το δίκτυο. Το δίκτυο όμως εις διάθεση όλων. Υπάρχουν διάφορες δυνατώσεις, ιδίως όσον αφορά τις ε, μεταφορές ταξιδιωτών. Ωραία, αυτό μια παρένθεση ήταν. Εδώ τώρα θα εξετάσουμε τη διάσταση πώς μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα και στις εμπαρευματικές μεταφορές στην Ευρώπη. Η κατανομή του ευρωπαϊκού συνδρομικού δικτύου σε διαδρόμους είναι σημαντική. Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί και μια τέτοια μεταφορά είναι σημαντικό ε, ε, εκείνοι που έχουν στα χέρια τους αυτά τα δίκτυα να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια μιας επιτροπής διαχείρισης όπως τόνισαν και ο κ. Μαρινέσκου και ο κ. Κράμερ. Ας πούμε αυτή τη διαδρομή Ρότερνταμ Τζένοβα που ανέφερε και ο κ. Κράμερ. Ένα one-stop shop <clears throat> δεν μπορεί να προγραμματίσει από μόνο του. Χρειάζεται πέντε επιχειρήσεις υποδομής. Το στην ε, ε, Ολλανδία, στην Γερμανία το Βέντε, στην ε, Ελβετία διαφορετικές επιχειρήσεις, ΕΣΠΕΤ, ΕΦΣΕΦΕΣ, τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις και στην Ιταλία Ρόμπο Φεροβίστα Τελεστάτο. Και θα πρέπει στην Επιτροπή αυτή τη διαχειριστική να συμφωνήσουν πότε μπορεί να περάσει αυτή η, μεταφορά. Ο καθένας έχει τη ο καθένας θέλει να κερδίσει κάτι. Πώς θα αποκλείσουμε δηλαδή το αναγνωριστικό με έναν one-stop ε, shop που καθορίζει από πού θα περάσει, πότε θα περάσει, πώς θα περάσει, γιατί θα περάσει. Ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Λοιπόν, για κάθε χώρα μία one-stop shop, όχι για κάθε διαδρομή, για κάθε χώρα. που θα καταγράφει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και θα έρθει σε επαφή με τους διαχειριστές της υποδομής όλων των λόγων δικτύων. Και αν υπάρχει μετά ένα πρόβλημα, Κάποιες χώρες έχουν παραδείγματος χάρη διαφορετικές ε, ράγες για τις εμπορευματικές μεταφορές. Εκεί όμως που συνδυάζονται και για τις εμπορευματικέ και τις ε, ε, ταξιδιωτικές μεταφορές κλπ. υπάρχουν προβλήματα. Και θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Και νομίζω συμφωνούμε ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα θα πρέπει το το δυνατό να επανέλθουμε στο κανονικό δρομολόγιο. Αυτό το one stop shop κατά τη γνώμη μου είναι πολύ χρήσιμο όταν συζητάμε σε παρεμποδίσεις σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν οι αιτήσει που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι δεν ε, πραγματοποιούνται μετά όπως θα έπρεπε. Τότε θα ε, πρέπει να έχουμε αυτό το one-stop shop σαν μια μονάδα διαιτησία. Στη Γερμανία έχουμε την Bundesnetzagentur, όπως τη λέμε, που κάνει ακριβώς αυτό που σας λέω, παίζει αυτό το ρόλο του one-stop shop θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και σε εμπορευματικέ μεταφορές. Δεν μπορούμε να πούμε εδώ έχει καθοριστεί αυτό και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από αυτήν ό,τι και να συμβεί. θα πρέπει να προγραμματίσουμε την χρήση κάθε διαδρομής αυτό το μοντέλο Rotterdam Rotterdam-Genova είναι με ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις εμπορευματικές μεταφορές και το παράδειγμα αυτό μπορούσε να μεταφερθεί μετά σε μεταφορές από την Ανατολή στη Δύση αλλά ο κάθε ε, ε ενδιαφερόμενος, ο κάθε ιδιοκτήτης υποδομής θα πρέπει να ξέρει Ωραία, εδώ έχουμε τώρα την προτεραιότητα των εμπορευματικών μεταφορών και θα συμφωνήσουμε ποια στιγμή θα τους δώσουμε δυνατότητα να μεταφερθούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Jā, um, uh, επειδή δεν είναι εδώ ο Σκιώδης που αντικαθιστώ, θα μιλήσω εγώ στη θέση του. Συμφωνώ ότι τα σημαντικότερα προβλήματα έχουν ταυτιστεί Πρέπει να βρούμε μια λύση ως προς αυτά με το Συμβούλιο και εγώ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το θέμα του καθεστώτος αυτού του one-stop shop. Παρακαλώ να ακούσουμε την επιχειρηματολογία του Συμβουλίου. Το θέμα δηλαδή είναι αν πρέπει πράγματι να δημιουργηθούν και νέα υπερεθνικά σώματα αν δεν έχουμε ένα καθαρό όραμα ή άποψη για το πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα, τότε να το ξανασκεφτούμε. Ίσως δεν πρέπει να δημιουργηθούν αυτά τα υπερεθνικά σώματα. Να, τα επιχειρήματα του Συμβουλίου είναι σοβαρά. Και δεύτερον, οι κατηγορίες των εμπορικών τρένων. Ίσως δεν πρέπει να είναι τόσο συγκεκριμένες και αυστηρές. Πρέπει γενικότερα να εκφράσουμε μερικές αρχές ως προς το πώς θα ταξινομούν ως προς τη χρήση των υποδομών αυτά τα εμπορευματικά τρένα. εξαρτάται και από, το, από την πυκνότητα της κυκλοφορίας. Παρακαλώ λοιπόν να είμαστε επικοδομητικοί. Μπαλζάιτης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαρινέσκου όπου πράγματι προσπάθησε να επιτύχει πολλούς συμβασμούς, ένα πολύ πολύ κείμενο. Δύσκολο είναι όχι μόνο για πολιτικούς, αλλά και για τεχνικούς λόγους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 20 διαφορετικά διαχειριστικά συστήματα για τις διαδρομικές μεταφορές και έχουμε και διαφορετικό πλάτος στις ράγες στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε πολλές δυνατότητε για να αυξήσουμε την το και να μειώσουμε τη μόλυνση. Γι' αυτό ο ρόλος των εμπορευματικών μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που δημιουργήθηκε ο λεγόμενος πρώτος κατάλογος που συμπεριλαμβάνει και κάποια σχέδια που ακόμα δεν είναι οικονομικά αποδοτικά αλλά που έχουν μια πολύ σημαντική προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που τελικά θα ε, δειχθούν και αποδοτικοί. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφορές ρωσικών αγαθών από την Αγία Πετρούπολη. Πετρούπολη. Θα μπορέσουν έτσι μεγάλες ποσότητες των μεταφορών να περάσει στους δρόμους και αυτό θα αυξήσει την αγωνιστικότητά μας. Πρόκειται σημαντικότητα της προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά κάποιον τρόπο στο μέλλον. Όσον αφορά αυτό το one-stop shop, Έχουμε διαφορετικά διαχειριστικά συστήματα και θα πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα πια. Κάτι σχετικά με το θέμα αυτό βέβαια. Δεν μπορούμε αμέσως να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε μια αρχή. Τώρα, όσον αφορά την ε, τροπολογία υπαριθμών 1, θα πρέπει βέβαια να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβασμό μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών. Και όσον αφορά τις προθεσμίες των δύο ετών που προβλέπονται στο κανονισμό, έχω να πω ότι βέβαια όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουν από την οικονομική κρίση. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη μας και δεν είναι ακόμα σαφές πότε θα βγουν από την κρίση όλες οι χώρες και αν. Γι' αυτό θα ήταν καλό να παρετείνουμε την προθεσμία αυτή σε πέντε χρόνια αντί δύο. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές απαιτούν όχι μόνο σημαντικές επενδύσεις, αλλά και σημαντικές προθεσμίες για μετατροπές. Κατά τα άλλα, συγχαίρω και πάλι τον εισηγητή. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voulais simplement dans la discussion nous rappeler. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώ να υπενθυμίσω ότι κατά την αποτίμηση της πρώτης ιδεροδρομικής δέσμης που γίνεται, νομίζω ότι 24 χώρες έχουν παραβιάσει τους ίδιους τους, τους κανόνες. Πρέπει λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη μας για, κατά τον συγγραφή αυτού του κανονισμού, γιατί δεν θα έχει νόημα να προβλέπετε κάτι αυστηρά εθνικό ή να προωθείται κάποιος, ε, κάποια συνδρομική εταιρεία η οποία παραβιάζει τους κανόνες. Όσο για το λεγόμενο one stop shop πρέπει να βρεθεί μια λύση για να μην υπάρχει υπερβολικό γραφειοκρατικό βάρος. Αυτό λένε οι εταιρείε μέχρι τώρα. Πρέπει να είναι κάτι αποτελεσματικός προς τη διαχείριση και των διαδρομών και της κυκλοφορίας γενικότερα και να προσφέρει κάτι. Νομίζω ότι ήδη ο κανονισμός δεν ήταν απολύτως απαραίτητος, αλλά αφού συζητιέται νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί κάποια εξισορρόπηση. Ο κανονισμός δηλαδή να προσφέρει κάτι στις υπάρχουσες εταιρείες και στις εμπορικές διαδρομές και να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι οι εθνικές υδροδρομικές εταιρείες παρεμποδίζουν, δεν θέλουν πιο ανεξάρτητη και καλύτερη διαχείριση κοινή. Αυτά τα τρία είναι τα κριτήρια και εγώ θα υπερψηφίσω οτιδήποτε επιτρέψει αυτή τη μεγαλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ εθνικών καθαρά συμφερόντων από τη μία και υπερβολικά συγκεντρωτικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών από την άλλη. Γιατί έτσι θα δυσκολέψουν τα πράγματα για όλους. Άι Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω κύριε Μαρουνέσκου για τα όσα κάνετε και να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές ε, για τη συνεργασία τους. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαρινέσκου κάτι το οποίο νομίζω ότι υπήρξε αντικείμενο από την αρχή το συζητή, από την αρχή. Το έθεσε και η κυρία Μπιλ για τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά για την απόφαση να τροποποιήσουμε και να συμπεριλάβουμε νέους ε, διαδρόμους. σε κάποιες περιπτώσεις, στη χώρα μας για παράδειγμα, υπάρχουν διάδρομοι ε, μεγάλης ταχύτητας ε, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κάποια στιγμή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κύριε Μαρινάσκου, στα άρθρα 3, 4 και 5 κυρίως, το Κοινοβούλιο δεν δέχεται επί της αρχής την κοινή θέση του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο ή με ποιον μηχανισμό έχουμε προβλέψει διότι από το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μου είναι σαφές τι μηχανισμό έχουμε προβλέψει για να τροποποιήσουμε λόγω διεύρυνθησης ή λόγω απαραίτητων αλλαγών διότι αν θέλετε αυτό δεν θα ολοκληρωθεί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια δυναμική διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο εμπορευμάτων και επιβατών ε, στην Ευρώπη. Τι μηχανισμό λοιπόν προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την μελλοντική εξέλιξη, να μην ε, έχουμε λοιπόν μια ε, διαδικασία ε, αυστηρή που κάνει μια τροποποίηση μια για πάντα. Τι μπορούμε να κάνουμε για βελτιώσει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κύριος Πασκουαρέλη. Συγγνώμη κύριε Πασκουαρέλη. Μάικολ, ήθελες να σχολιάσεις κάτι. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, κύριε Κούν, στη Γερμανία. Οι εθνικέ επιχειρήσεις παίρνουν εθνικές ε, ε, επιδοτήσει για τα εθνικά δίκτυα. Αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο θέλει, αλλά οι ιδιώτες δεν παίρνουν καμία ενίσχυση για την συντήρηση των δικτύων αυτών. Είναι αναγκασμένοι δηλαδή από τις εισπράξεις του να κάνουν τη συντήρηση και την εξέλιξη. Αυτό εννοούσε προηγουμένω. Υπάρχουν διαφορές, προσπαθούμε και με τη νέα κυβέρνηση κάτι να πετύχουμε, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ ιδιωτικών δικτύων και κρατικών. Okay, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πασκουαρέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω εξ ονόματος της Κομισιόν ότι αναγνωρίζουμε την εργασία του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ΜΕΤΑΦ δηλαδή. Ιδιαίτερα σε αυτήν τη θητεία με τον κύριο Μαρινέσκου. Καταλήξαμε σε μια κοινή θέση, το Συμβούλιο κατέληξε μια κοινή θέση αρκετά επικοδομητική και Γι' αυτόν τον λόγο τη δέχτηκε και η Κομισιόν. Αλλά επί τεσσάρων σημείων αρνείται τις καινοτομίες που προτείνουμε. Αντίθετα έχει υποβάλει μία τροπολογία που λέει ότι σε αυτόν τον κανονισμό τίποτα δεν πρέπει να αλλάζει την υπάρχουσα νομοθεσία. Είναι λοιπόν ένας πολύ σοβαρός αυτοπεριορισμός που επιβάλλει το Συμβούλιο εναντίον όλων των καινοτομιών του κειμένου. Και αυτά τα τέσσερα σημεία είναι αυτά που ανέφερε ο κύριος Μαρινέσκο, το One Stop Shop, που δεν είναι καθόλου κάτι το καινούριο ή ένα και νέο πυρεθνικό σώμα που υπόθηκε κτλ. Είναι απλώς ένα εργαλείο για να λειτουργήσουν καλύτερα οι διάδρομοι ή οι διαδρομές γιατί πρόκειται εδώ για λειτουργική συνεργασία μεταξύ υπαρχουσών υποδομών, δηλαδή σιδηροδρομικών εταιριών. Υπάρχει ήδη το RailNet Europe με έδρα τη Βιέννη που έχει εφαρμόσει ήδη το One Stop Shop για να κλείνει διαδρομές. Και αυτό το One Stop Shop λοιπόν, όσο και να λέει το RailNet αυτό, δεν είναι καινοτομία καθόλου. Απλώς υποβάλλει, μεταφέρει αιτήματα διαδρομών στους ενδιαφερόμενους και μέχρι τώρα αυτό το One Stop Shop της Βιέννης δεν είναι πολύ αποτελεσματικό γιατί καλύπτει μόνο το 5% των αιτημάτων για νέες διαδρομές. Είναι λοιπόν σύστημα που δεν δουλεύει και η δική μας πρόταση θέλει να δουλέψει. Δεν πρόκειται λοιπόν επαναλαμβάνω για κανένα νέο οργανισμό της Ένωσης αλλά για ένα ολόκληρο καινούργιο εργαλείο που να έχει κάποια πιο αυτόνομη ευθύνη. Αυτόνομη δεν σημαίνει τελείως ανεξάρτητη και χωρίς καμία σχέση με τους υπάρχοντες εθνικούς κανόνες, όχι, Έπειτα, οι λεγόμενοι authorized applicants. Για μας αυτό είναι κάτι που διευκολύνει τη διευθέτηση του ανταγωνισμού, δηλαδή. Ε? Αν κάποιοι που δεν είναι συνδρομικές εταιρείε έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από διάφορες σιδηροδρομικές εταιρείες που υπάρχουν στην αγορά να μας κάνουν μια προσφορά τιμών για να διαλέξουν την πιο συμφέρουσα προσφορά, ε, τότε αυτό το σύστημα του authorized applicant νομίζω ότι είναι κάτι το σωστό γιατί αφήνει στο κάθε κράτος τη δυνατότητα να κάνει κάτι που δεν υπάρχει στο έθνος αυτό. Τρίτο σημείο. Οι κανόνες προτεραιότητας. Και εδώ να μην παρεξηγηθεί αυτό που είπαμε. Εμείς δεν προτείνουμε τα εμπορευματικά τρένα να έχουν πάντα προτεραιότητα ενώ τα επιβατικά και τα ποστάλια να χρειάζονται πάντοτε να περιμένουν για να περάσουν πρώτα τα εμπορεύματα. Όχι καθόλου μάλιστα, καθόλου. Απλώς δεν θέλουμε άνηση μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων τύπων μεταφοράς. Να υπάρξουν κοινοί κανόνες. Δεν θα τους καθορίσει η Κομισιόν και η Ένωση, αλλά οι ίδιοι διαχειριστές των σιδηροδρομικών εταιριών, που τώρα τους λέμε των υποδομών. Λοιπόν, τέταρτο σημείο, η governance των διαδρόμων θέλουμε και εδώ να υπάρξει ένας οργανισμός ας πούμε κάποιο γκρουπ οικονομικών συμφερόντων ή υποδομών που να μην είναι απλώς ένα talking shop μια συνάντηση φίλων που να κάνουν κουβεντούλες δηλαδή αλλά να μπορεί να κάνει επενδύσεις να διαχειρίζεται τις υποδομές για να είναι πιο ρέουσα η κυκλοφορία. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία όπου το Συμβούλιο αρνείται και θέλει να παραμείνουν τα πράγματα όσοι έχουν. Και όπως είπε και η κυρία Ντουράν, εδώ πρέπει να βρεθεί κάποια εξισορρόπηση, να γίνουν αμοιβέ υποχωρήσει. γιατί αν υπάρχει συμφωνία επί αυτών των τεσσάρων σημείων θα πετύχουμε. Ή θα αποτύχουμε. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που θα μπορούσα να αναφέρω αλλά προτιμώ να μην το κάνω μεταξύ των οποίων είναι και η επιλογή των διαδρόμων ή διαδρομών. Η Κομισιόν δέχεται συμβιβασμό επί της κοινή θέσης. Οι διάδρομοι δηλαδή που έχουν επιλογή είναι εννέα. Έξι από αυτούς ανταποκρίνονται σε διαδρόμους RTMS που ήδη έχουν λάβει το κοινοτικό βάπτισμα και από τους οποίους οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύουν παρά 6% σε χιλιόμετρα αλλά 20% της κυκλοφορίας. Βλέπετε πόσο σημαντική είναι και πόσο λογική είναι αυτή η επιλογή επομένως. Οι τρεις υπόλοιποι διάδρομοι είναι διάδρομοι επί των οποίων οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν απολύτως. Οι παράγοντες δηλαδή. Έχουν καθοριστεί από εκείνον τον οργανισμό που σας ανέφερα προηγουμένως της Βιέννης Real Αν λοιπόν Συμβούλιο και Κενοβούλιο μαζί με μας θέλουμε έναν ευρωπαϊκό συντηροδρομικό χώρο, ολοκληρωμένο όμως, ολοκληρωμένο, και που να βασίζεται στους νενομημένους <clears throat> διαδρόμους, για να γίνει αυτό δεν αρκεί να ε, βάλουμε τα υπάρχοντα, τους υπάρχοντες διαδρόμους και να προσθέσουμε σε αυτούς τους καινούριους. Πρέπει να υπάρξουν δομές λήψης αποφάσεων πιο ολοκληρωμένες, να δούμε ποιοι θα είναι οι νομισμένοι ετούντες κτλ. Η κυρία Ντουράν είπε ότι ίσως να μην χρειάζεται καν κανονισμός για να διαθετηθούν όλα αυτά, αλλά η Κομισιόν είπε επανειλημμένα ότι ο κανονισμός χρειάζεται. Είναι κάτι το προφανές για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος. Αφού ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα σχετικό εθνικά από τους incumbents, δηλαδή τις εθνικές σιδηροδρομικές εταιρείες. Τώρα τις λέμε incumbents. και οι διαχειριστές των υποδομών, δηλαδή οι διευθυντές των υποδομικών επιχειρήσεων, εταιριών, δεν αρκούν για να τα λύσουν όλα αυτά. Λοιπόν, αφού θέλουμε καινοτομίε, πρέπει να βρούμε λύσει επί των τεσσάρων αυτών προβλημάτων που ανέφερε και ο κύριο Μαρινέσκου. Αυτέ είναι οι απαραίτητε προποθέσει για να υπάρξει ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο όπου η κυκλοφορία των εμπορευμάτων να μπορέσει να ανθίσει σιδηροδρομικά εφόσον βέβαια θέλουμε να υποκαταστήσει τις οδικές μεταφορές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρινέσκου μήπως, γιατί ξέρω ότι από αυτά που είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ θα θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Πρώτον, μία γενική δήλωση. Όταν νομοθετούμε πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτόμαστε τι προσφέρει αυτή η νομοθεσία. Γιατί άμα δεν το ξέρουμε αυτό τότε δεν έχει κανένα νόημα να νομοθετήσουμε. Λοιπόν, για τους εμπορευματικούς διαδρόμους, γιατί ζητούμε διευθέτηση. Για να βελτιώσουμε τα κακό κείμενα. Και ποια είναι αυτά. Πρώτον, λείπει συντονισμός. Διότι υπάρχουν εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές, υπάρχουν και άλλα συστήματα η RTMS, RailNet Europe και άλλα. Υπάρχουν λοιπόν άλλες επιλογές, αλλά δεν υπάρχει συντονισμός των, της κυκλοφορίας στους εμπορευματικούς αυτούς διαδρόμους. Δεν υπάρχει λοιπόν συντονισμός για να μπορεί ένα εμπορευματικό τρένο να κυκλοφορήσει θεωρητικά όπως τα επιβατικά. Διότι πιστεύω ότι από τεχνικής απόψεως υπάρχει τεχνική δυνατότητα δυνατότητα λέγω να μπορεί ένα τρένο να φεύγει από τη Γένοβα και να φτάνει μέχρι το Ρότερνταμ χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Σαν επιβατικό δηλαδή. Τεχνικά γίνεται, αλλά για να επιτευχθεί αυτό που τεχνικά γίνεται χρειάζεται συντονισμός. Ο κανονισμός λοιπόν αυτό στοχεύει ακριβώς στη βελτίωση του συντονισμού, δηλαδή Πρώτον, με τη διευκόλυνση αυτή των εμπορευματικών μεταφορών γιατί, που έχει διάφορα ονόματα από διάφορους παράγοντες και τα τρία θεσμικά όργανα όμως συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει ο συντονισμός δεύτερον το One Stop Shop που δεν είναι όργανο όπως είπε κάποιο και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Είναι μια υπηρεσία όπου μπορεί να υποβληθεί μια αίτηση και η υπηρεσία θα συνεργάζεται με, τις υπάρχο, με τα υπάρχοντα με τις υπάρχουσες εθνικές εταιρείες γιατί αλλιώς δεν γίνεται και μετά το One Stop Shop θα δε βλέπει αν το γαλλικό, η γαλλική ας πούμε εταιρεία έχει εμποδίσει ένα γερμανικό τρένο να περάσει από τη Γαλλία για λόγους μη τεχνικούς. Να μπορεί να το ελέγξει αυτό. Και έτσι μόνο θα είμαστε βέβαιοι ότι οι εθνικές εταιρείες και οι εθνικές υπηρεσίες συντονισμού των σιδηροδρόμων θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ικανοποιήσουν τους ετούντες. Αυτή είναι η ιδέα του One Stop Shop. Ξέρω ότι σας έχουν πλησιάσει και πιέσει εκπρόσωποι των σιδηροδρομικών εταιριών. Εκείνοι είναι αυτοί που αντιτίθενται στην εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος γιατί εκείνοι θεωρούν ότι θα χάσουν τον έλεγχο της αγοράς. Πρέπει όμως εδώ να υπάρξει καινοτομία. Δηλαδή καλύτερη governance γιατί αυτή η διαχειριστική επιτροπή που είπαμε πληρεί και ένα άλλο κριτήριο, δηλαδή διευκολύνει τις επενδύσεις στις υποδομές. Αυτή η διαχειριστική επιτροπή θα συντονίζει και τις επενδύσεις πάνω στον ίδιο διάδρομο διαφορετικές επενδύσεις στον ίδιο διάδρομο. Άρα θα διευκολύνονται οι επενδύσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι το One Stop Shop πρέπει να εισαχθεί, να εφαρμοστεί. Και μετά τις πρώτες συζητήσεις μας με το Συμβούλιο νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει. Στη δε προσθήκη ή παράρτημα που, στην οποία έχουν αναφερθεί πολλοί, το παράρτημα 1. Στην αρχική πρόταση της Κομισιόν έλεγε ότι μέσα σε τρία χρόνια, αν δεν απατώμε, σε τρία χρόνια, κάθε χώρα μέλος θα είναι μέρος ενός διαδρόμου και αυτό υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Εάν υπάρχει βέβαια σιδηροδρομική σύνδεση με τις άλλες χώρες του διαδρόμου. Το Συμβούλιο λοιπόν έκανε μια πρόταση πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή, ότι δηλαδή ο κανονισμός αυτός να αποφασίζει και για τους πρώτους νέους διαδρόμους. Αυτό καλό είναι. Γιατί πρέπει να καθοριστούν αυτοί οι πρώτοι διάδρομοι χωρίς να περιμένουμε τρία χρόνια μέχρι να αποφασίσει το κάθε κράτος μέλος λοιπά. Τώρα, από ποιες χώρες περνάνε οι διάδρομοι αυτοί, εγώ πρότεινα να γίνει μια ειδική συνεδρίαση μόνο και μόνο για αυτό το θέμα στο παράρτημα 1. Να συζητήσουμε πρώτα την ουσία του κανονισμού και μετά χωριστά τις λεπατομέρειες που από πού θα περνάνε οι διάδρομοι και τα λοιπά. Γιατί το θέμα της Ισπανίας τώρα εκεί έχει δύο διαδρόμους και κατ' εμέ είναι οι μόνοι διάδρομοι που μπορούν να υπάρξουν στην Ισπανία. Περνάνε και από τη Γαλλία βέβαια προφανώς. Αλλά υπάρχει ίσως η δυνατότητα να ζητηθούν και αλλαγές. Και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καθορίσει με ποια κριτήρια προτείνονται οι διάδρομοι αυτοί. Το ζητήσαμε ήδη, περιμένουμε την απάντηση, αλλά ξέρουμε ήδη ότι το παράρτημα αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μέλη πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν σε τουλάχιστον ένα διάδρομο μέσα σε τρία χρόνια. Υποχρεωτικά. Να μην σπαταλήσουμε κι άλλο χρόνο γι' αυτό, αλλά να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Τώρα, πώς θα μπορούσε να αλλάξει το παράρτημα να τροποποιηθεί. Το παράρτημα αυτό, το ένα δηλαδή, παράρτημα 1, λέει ότι οι πρώτοι διάδρομοι δεν μπορούν να αλλάξουν. Αφού είναι οι πρώτοι, πώς θα αλλάξουν. Οι χώρες μέλη όμως, το λέει αυτό ο κανονισμός, οι χώρες μέλη μπορούν να προτείνουν εναλλακτικού διαδρόμους ή να αλλάξουν τους υπάρχοντες που δεν μπορούν να αλλάξουν. Η Κομισιόν θα τα αποφασίσει αυτά η Κομισιόν. Ο κανονισμός το λέει και αυτό το λέει. Θα το αποφασίσουν οι χώρες μέλη αλλά η Κομισιόν θα το καθορίσει. Το λέει ο κανονισμός. Λοιπόν, τα κριτήρια δηλαδή για τις αλλαγές για τη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου. Τα κριτήρια. Και το λέει ο κανονισμός, το επαναλαμβάνω. Υπάρχει τρόπος πρότασης νέων διαδρόμων ή διαδρομών. Το λέει μέσα το λέει. Στο άρθρο 3, στο σημείο 3 για την κοινή διαδικασία, στη δική μου πρόταση λέω τώρα, στη δική μου πρόταση, το σημείο 3 μιλάει για την κανονική διαδικασία, πώς υποβάλλει κανείς αίτηση για να εγκριθεί ένας διάδρομος, ενώ το σημείο 4 αφορά το παράρτημα και μόνο το παράρτημα. Κατά τα υπόλοιπα, σας το είπα ήδη, μπορούμε να κάνουμε μια, μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμό με το, πώς να το πω, με το Συμβούλιο, Συμβούλιο, που να αλλάζει την περίοδο τριετή, πενταετή, δηλαδή Μέσα λέω στον κανονισμό το λέει. Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας διάδρομος. Τι θα πει αυτό να ενεργοποιηθεί. Να υπάρχει one stop shop και διαχειριστική επιτροπή. Γιατί να χρειάζονται πέντε χρόνια γι' αυτό. Για να ενεργοποιηθεί ο διάδρομος. Δεν χρειάζονται πέντε χρόνια. Είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Και για τους πρώτους τουλάχιστον διαδρόμους αρκούν νομίζω δύο χρόνια χωρίς πρόβλημα. Γιατί αυτά αρκούν για να υπάρξει ένας διάδρομος και να λειτουργήσει. Και μετά βέβαια για τις επενδύσεις αυτό είναι άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ σας, ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκο. Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε είναι προθεσμένη την υποβολή των 12 Απριλίου η εξέταση των τροπολογιών στην Επιτροπή Μεταφορών 3 Μαΐου, ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών 4 Μαΐου και ελπίζουμε να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Ωραία. Λοιπόν, 12 Απριλίου προθεσμία την των τροπολογιών. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου για την παρουσίαση αυτή, την τόσο λεπτομερή. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Ράνα για τους κοινωνικούς κατώνες στις οδικές μεταφορές. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων, κύριε Ράνο, που δεχτήκατε να τεθεί αυτό το θέμα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε περισσότερο χρόνο για την Ισπανική Προεδρία το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την ε, ευελιξία σας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ καταρχήν να επανέλθω στη συζήτηση του εγγράφου εργασία. Έχουμε μπροστά μας σήμερα μια πρόταση ε, έκθεσης που προσπάθησα να συγκεντρώσω στις κοινωνικούς κανόνες τις οδικές μεταφορές και να σας πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα το ύψους των κυρώσεων, αλλά και η ταξινόμηση των διαφόρων ε, παραβάσεων. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για ένα διαμεθοριακό πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στην οικονομία μας που πλήττονται από αυτό. Διακόπτει ο πρόεδρος, μη συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Μαρινέσκου, προσπαθώ να βλέπω την επόμενη συγκήτρια και δεν μπορώ γιατί έχετε κάποιο πηγαδάκι εκεί και δεν βλέπω την κυρία Ράνερ που είναι πίσω σας. Παρακαλώ, όποιος θέλει να συναντηθεί με τους συναδέλφους να βγει από την αίθουσα. Η κυρία Ράνερ, ναι, ναι. Ξέρω ότι το προηγούμενο θέμα ήταν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά νομίζω ότι και το δικό μου θέμα δεν είναι τόσο μικρή σημασία. Και ελπίζω να παραμείνουν κάποιοι συνάδελφοι στην αίθουσα. Θα είμαι βέβαια σύντομη γιατί πρόκειται για την απαρχή τη συζήτηση ένα αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να βασίζεται μόνο σε διαφανεί και συγκρίσιμες κυρώσεις. Σε σχέση με την προετοιμασία της ε, έκθεσης είχα πάρα πολλές ε, συζητήσεις και με μεταφορικές επιχειρήσεις αλλά και με οργανώσεις εργαζομένων και εκπροσώπους κάποιων κρατών μελών. Και ε, είδα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα ως νομικό Κατανοητό βέβαια ότι τα συστήματα κυρώσεων στα διάφορα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ διαφορετικά και βασίζονται ιστορικά σε διαφορετικά νομικά συστήματα και διαφορετικά οικονομικά συστήματα. Διακόπτω πρόεδρος, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κύριε Μαρινέσκου, κύριε Γιάλα Σέντα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, είναι σημαντικό, το ξέρω. Αλλά δεν είναι σωστό για την κυρία Ράνα αυτό που κάνετε ελπίζω να υπάρχουν παρόμοιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις και για τη δική μου έκθεση. Λοιπόν, έλεγα ότι αν συζητήσει κανένας με τους ότι χρειάζεται να δράσουμε. Βέβαια, υπάρχει το θέμα και πρόβλημα της επικουρικότητας και του παρέμβαση στα εθνικά συμφέροντα. Αλλά λόγω της ε, οδικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη καλύτερη παρακολούθηση, καλύτερος έλεγχος θα έλεγα. Δεν μπορούμε από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους εφόσον δεν υπάρχουν και σχετικοί έλεγχοι. Και περαιτέρω, επίσης σημαντικό για ένα πρώτο βήμα, η έλεγχοι αυτή και τα αποτελέσματα των κυρώσεων να ε, κοινοποιούνται αμοιβαία στα κράτη-μέλη. Και επ' αυτού προτείνω να υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για Στατικές Μεταφορές που θα συντονίζει αυτό το έργο. Εάν εγώ ως κρατοσμένος δεν ξέρω ποιε είναι η κύρωση σε μια άλλη χώρα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεταφορές δεν γίνονται από μία χώρα στην άλλη μόνο, αλλά μέσω τριών, 4, 5, 6 χωρών. Εγώ θα πρέπει λοιπόν ως επιχειρηματίας να γνωρίζω ποιε είναι οι διατάξεις σε κάθε ε, κράτος που θα πρέπει να τηρούνται από τα οχήματά μου. Καμιά φορά υπάρχουν κάποιες διατάξεις που δεν τηρούν και αντιμετωπίζονται διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη λόγω της αρχής επικουρικότητας. Επίσης, θα μπορούσαμε επίση να σκεφτούμε και το εξή. Το άρθρο 83 παράγραφος της συνθήκης της Λισαβόνας θα μας έδινε τη δυνατότητα για μεγαλύτερη παρέμβαση εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητα αναγκαίο. εξέτασα προκαταρτικά τη δυνατότητα αυτή και με τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτρες και ελπίζω ότι όταν υπάρχει τώρα η έκθεση γραπτά θα μπορέσουμε να επισέρθουμε σε αυτή. Δεν ήταν ακόμα επαρκή η συζήτηση με τους σκιώδεις, ήταν μονάχα μια προκαταρτική συζήτηση που θεωρούσα απαραίτητη για να μπορούσαμε να περάσουμε τώρα στις έντονες συζητήσεις και να συλλέξουμε τις απόψεις και των άλλων συναδέλφων. Χαίρομαι να του ακούσω, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχουν ε, να πούνε και αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε διαφορετικέ απόψει και να μην πετύχουμε μία ενιαία άποψη. Μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ μόνο αν πετύχουμε ομοφωνία εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών και το ελπίζω πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αλκατράουη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Διότι άλλο είναι να ε, ψηφίζει κάποιος νομοθεσία και άλλο είναι να δούμε πώς υλοποιείται. Οι στόχοι μας, οι οποίοι καθορίστηκαν αρχικώς, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον επετέχθησαν. Βάσει και τις συζήτηση που είχαμε κάνει στο παρελθόν, ε, προέκυψε το κείμενο τη εισηγήτρια, το οποίο διαπιστώνει ότι υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία μας το υπενθυμίζουν. Όπως είπα λοιπόν είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Κάποιες προτάσεις τις οποίες θα ήθελα να κάνω εξ ονόματος ομάδος μας. Συμφωνούμε με το κεντρικό μήνυμα της εισηγήτριας, δηλαδή ότι είναι απαραίτητη περισσότερη εναρμόνιση όσον αφορά στις κυρώσεις η εισηγήτρια δικαίω λέει ότι βάσει και τη συνθήκη Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νέε νέες δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον οι προσανατολισμοί μας ε, μπορεί να είναι ε, πιο δεσμευτικοί. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και σχετικές προτάσεις. Όσον αφορά τώρα την εκτέλεση, την υλοποίηση. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε ε, κατά πόσον υπάρχουν έλεγχοι, κυρίως την έλεγχη στα αυτοκίνητα οχήματα. Ε, όσον αφορά τώρα τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ε, το είπαμε και στη συζήτηση για την έκθεση Gross, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να γίνει και μια εις βάθος ανάλυση προηγουμένως. Θα πρέπει να συζητήσουμε δηλαδή την χρησιμότητα, την ανάγκη μιας τέτοιας υπηρεσίας ε, τι αρμοδιότητες θα έχει, τι πόρους θα διαθέτει η υπηρεσία αυτή και να δούμε κατά πόσον θα υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία για αυτή την υπηρεσία. Διαπιστώνω ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετές ιδέες για τις αρμοδιότητες αυτής της ε, υπηρεσίας μας, της η συγγήτρια Αναφερόμαστε σε ελάχιστο κανόνες κατάρτισης ε, για τους αρμόδιους υπαλλήλους. για στατιστικά στοιχεία, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να συστηθεί μια νέα υπηρεσία. Μπορεί να το κάνει κάλλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνει μια συζήτηση για την υπηρεσία αυτή για να δούμε κατά πόσον μας χρειάζεται. Ολοκληρώνοντας όσον αφορά στην ε, κοινοποίηση, ε, να υπάρχει επικοινωνία για τα βαρέα οχήματα, επί παραδείγματα, υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές στην εφαρμογή και δεδομένου ότι υπάρχουν και αρκετές νομοθετικές πράξεις για το θέμα αυτό, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ίσως και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, να έχουμε ε, μια μορφή πηξίδας αν θέλετε, π.χ. το GPS. Γιατί να μην μπορούμε να έχουμε αυτές τις πληροφορίες ε, και σε εθνικό επίπεδο για τους οδηγούς θα πρέπει κάπως να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες. Θα σταματήσω εδώ. Ε, σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε με την εισηγήτρια στα βασικά σημεία και από εκεί και πέρα θα δούμε τι τροπολογίες μπορούμε να καταθέσουμε προκειμένου να διευκρινίσουμε κάποιες πτυχές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Μέσνερ. Δυστυχώ, ο, ο σχεδόν ηγητή της ομάδας μας κ. Στραμάζα απουσιάζει. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Ράνιν για την καλή συνεργασία και εξ ονόματο του εισηγητή. Θα υπάρχουν και μελλοντικέ συζητήσει με του κοιόδε. Εγώ εξ ονόματο τη ομάδα έχω να σα πω απλώ ότι υπάρχουν ήδη μια σειρά κανόνων που υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τηρούνται, κατά πόσο τηρούνται σωστά. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσουμε στα πλαίσια αυτής της οδηγία για τις κοινωνικέ διατάξεις των οδικών μεταφορών και μετά να δούμε ε, τι γίνεται σχετικά με το χρόνο ανάπαυσης των οδηγών κατά πόσον όταν προβλέπουμε εμεί συγκεκριμένου όρου ανάπαυσης και συγκεκριμένου διάρκεια οδήγηση, αν υπάρχουν παραδείγματο χάρη αρκετά, αρκετά πάρκινγκ για να μπορέσουν τα φορτηγά αυτά να σταθούν. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε αφενό να προωθήσουμε την οδική ασφάλεια, από την άλλη μεριά να μην επιβάλλουμε υπερβολική γραφειοκρατία που θα περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερα. Αν υπάρχουν δυνατότητε απλούστευση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Θα παρακολουθούσα με ενδιαφέρον την συνέχιση τη συζήτηση και την επόμενη φορά σα λέω θα είναι παρόν και ο κύριο Τρεμόζα οπωσδήποτε και θα είναι και παρόν και στι επιμέρου συζητήσει με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την εργασία της. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι ένα θέμα πολύ γνωστό εδώ στην Επιτροπή μας είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε των σημαντικών σημείων το λιγότερο δυνατόν θα έλεγα. Κατά μένα παραμένουν δύο σημεία ανοιχτά, σημαντικά σημεία για το θέμα. Καταρχήν θα πρέπει οριστικά να συμφωνήσουμε τι ε, θεωρείται στα διάφορα κρατημέρια ε, πολύ σοβαρή παράβαση, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, να εξάσουμε το θέμα της συχνότητας των ελέγχων. Αυτό το θέμα της συχνότητας των ελέγχων, κατά με, παραμένει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί όταν ξέρουμε ότι σε ορισμένε χώρες ο έλεγχος είναι κάτω από το 2%, τότε η αρχή της επικουρικότητας ε, δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε τα κράτη-μέλη, αλλά πρόκειται για ένα επικίνδυνο όπλο να μην γίνονται κάποιοι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν. Όσον αφορά τις καταυστές τις ε, κυρώσεις, ξέρουμε ότι διαφορετικού ύψους, διαφορετικής ε, διαβάθμισης δεν είναι προσαρμοσμένες, είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Ε, στη περιοχή στην οποία ζω εγώ, αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα και διαφορές. Δηλαδή σε μια χώρα αποσύρεται η αδειοδήγηση, και θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα οδήγησης από μια χώρα η οποία δεν είχε εκδώσει καταρχήν την άδεια οδήγηση κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδίω ε, στον χώρο αυτών προσαρμοσμένων δυνατοτήτων. Το ένα είναι θέμα της συνεννόησης, το δεύτερο είναι το θέμα της ε, ε οικονομικής αποδοτήσης των επιχειρήσεων, το τρίτο είναι η ασφάλεια των ε, παθητικά και ενεργικά συμμετοχών στις οδικές ε, μεταφορές. Και τέλος ε, το θέμα ότι η επικουρικότητα θα πρέπει να παίζει μικρότερο ρόλο τα πρόκειται για θέματα ασφάλειας. Ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστούμε κύριος Μπράτμπορν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω αν ανατρέξουμε όπως είπε και η κυρία Ράνερ στην πρώτη συζήτηση που κάναμε επί του θέματος εγώ τότε είχα πει ότι το σκεπτικό είναι καλό, αλλά με όλες αυτές τις διάφορες μορφές νομοθεσίας, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και τότε είχα πει ότι αυτά τα προβλήματα δεν ε, λύνονται με μια ενέα αντιμετώπιση για όλα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ε, το 2% μόνο είναι διαμεθοριακές ε, μεταφορές εμπορικές. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην ε, ε, υπόλοιπη Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις και το επεσήμανε και ο κύριος Γκρός και η κυρία Λίχτεμπεργκερ σε προηγούμενη περίπτωση αναφέρθηκε στο πρόβλημα της Αυστρίας. Καταλαβαίνω ότι ανησυχίες υπάρχουν εκεί. Αλλά για μένα η όλη προσέγγιση, ε, ο βασικός όρος θα πρέπει να είναι επικουρικότητα. Να σταθώ τώρα σε κάποια σημεία της έκθεσης κυρία Ράνερ. Ε, νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσει κύριε Πρόεδρε το γεγονός ότι δεν θα διατρέξω την έκθεση ε, ανά σημείο, ε, διότι συμφωνώ με κάποια σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να περιοριστώ σε κάποιους βασικούς και μόνον τομείς. Πρώτον, η κυρία Ράνερ ζητά μία υπηρεσία οδικών μεταφορών και ο κύριος ε, ε, ε, Αλκαντράου είπε ότι πρέπει να το συζητήσουμε κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε, θα θυμάστε ότι στην τελευταία θητεία του Κοινοβουλίου και νομίζω και στην προτελευταία θητεία συνεχώς συζητούσαμε κατά πόσον χρειαζόμαστε μια υπηρεσία για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και η απάντηση ήταν πάντα όχι. Εγώ δεν έχω αλλάξει άποψη για το κατά πόσον χρειαζόμαστε λοιπόν μια υπηρεσία οδικών μεταφορών και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες υπηρεσίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ε, στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Δείτε τι χαμό ε, έχουν δημιουργήσει αυτές οι υπηρεσίες. δίνουμε χρήματα ε, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με λαθασμένο τρόπο αν δημιουργήσουμε μια τέτοια υπηρεσία. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση. Η δεύτερη παρατηρήσή μου είναι το θέμα της προσέγγισης με το ποινικό δίκαιο. Στην προηγούμενη θητεία, ευτυχώς ή δυστυχώς, ήμουνα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που συζητούσε την ε, λεγόμενη προσέγγιση του ποινικού δικαίου. Ε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αναρμόνιση του ποινικού δικαίου. Και πάλι διαπιστώνουμε ότι στο κείμενο αυτό υπάρχει μια αντίστοιχη πρόταση. Αυτό το οποίο διαπιστώνω εγώ πάντα σε οποιαδήποτε απόπειρα εναρμόνισης ποινικού δικαίου είναι ότι το κάθε κράτος μέλος ε, για ιστορικούς λόγους έχει διαφορετικά νομικά συστήματα και το δικό μου και το δικό σας ε, κύριε Πρόεδρε αλλά και στις άλλες ε, χώρες ακολουθείται μια τελείως διαφορετική νομική πρακτική. Η απόπειρα λοιπόν να εναρμονίσουμε το ποινικό δίκαιο στον τομέα αυτό όχι μόνο θα ήταν αντιπαραγωγική αλλά δεν είναι και επιθυμητή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ε, μου το επεσήμαναν εμένα και φαντάζομαι ότι θα το επεσήμαναν και σε εσά κύριε Πρόεδρε. Παραδείγματο χάρη, για ε, παραβιάσεις ε, κυκλοφορίας δεν υπάρχει ποινική διαδικασία. Ε, δεν υπάρχει διαδικασία έφεση. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή αποφασίσουν ότι κάποιο είναι ένοχο, δεν υπάρχει διαδικασία έφεση. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αντιβαίνει στην έννοια της ε, δίκαιης και αμερόληπτης δικαιοσύνης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η εναρμόνιση ποινικού δικαίου θα είναι αποτελεσματική στον τομέα αυτό. Και αυτό παραβλέποντας και τις όλες παραδόσεις του τι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν πολύ σοβαρά οδικά παραπτώματα και κάποιοι άλλοι όχι. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα αυτών των πρακτικών σήμερα και δεν θα μπορούσα να δεχτώ και την ε, παρατήρηση του κυρίου Αλκαντράουι, την εισαγωγή της τεχνολογίας και του GPS για να ε, εντοπίζει κανείς όλα τα εμπορικά οχήματα. Μιλάμε για μεγάλο αδελφό εδώ και φυσικά αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν θα ήθελα να τελειώσω με αρνητικό τρόπο, θα ήθελα να τελειώσω με κάτι θετικό. Ως προς τις άλλες πρωτοβουλίες που προτείνει η κυρία Ραν στην έκθεσή, του, την έκθεσή της, στην παράγραφο 21 για παράδειγμα αναφέρεται στην κατάλληλη υποδομή για να συνδράμουμε τους οδηγούς και όπως γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή εξέταζε την ιδέα των ασφαλών μέσων ε, και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε στις πτυχές της ασφάλειας αυτών των εγκαταστάσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε στην ασφάλεια και με τους δύο τρόπους. Νομίζω ότι τα προβλήματα που έχουμε δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων που ε, κάνουν οποιαδήποτε παραβίαση, αλλά το γεγονός ότι η εμπορική κυκλοφορία σε μεγάλα λιμάνια, για παράδειγμα, εξακολουθεί να γίνεται τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στην ε, ε, ασφάλεια, λοιπόν, ε, με τη μία έννοια, αλλά και με τις δύο έννοιες, τη χρήση των οδικών οδών και ούτω καθεξής. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μπορεί αυτό το πρόβλημα να ανακύπτει συνεχώς ε, και επειδή στα γαλλικά οι όροι safety και security είναι αντίστροφοι, δεν ξέρω πώ μπορεί να τα συμπεριλάβει αυτά η εισηγήτρια. Έχω τρει ακόμα μιλητέ. Ο κύριο Κράμερ. Η κυρία Λιχτεμπέργκερ δεν είναι εδώ είναι σε κάποια άλλη επιτροπή όπου πρέπει να παρέμβει και να ψηφίσει, επομένω δεν μπορεί να είναι παρούσα. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια εξ ονόματο τη. Θα σταθώ σε τρεις πτυχές. Ε, η υπηρεσία οδικών μεταφορών. Δεν ξέρω γιατί είναι απαραίτητη μια τέτοια υπηρεσία. Υπάρχουν τεχνικοί κανόνες, ενισχύ, που πολύ συχνά ε, επικρίνονται κιόλας, αλλά η υπηρεσία δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Αυτό όμως που χρειαζόμαστε είναι θέλουμε να φροντίσουμε οι κανόνες να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, να είναι συμβατοί, να μην είναι διαφορετικοί και να μπορούν πολύ πιο γλίγορα να ε, ε, ε, ορίζονται. Στην Ελβετία, παραδείγματο χάρη, να παρόν, όταν έγινε ένας έλεγχος ενός φορτηγού, αλλά για να βρουν όλα τα στοιχεία διαρκούσε πάρα πάρα πολλές ώρες. Και οι, οδηγοί θέλουν να ελεγχθούν, γιατί ε, ε, υποχρεώνουν από τους εργοδότες τους να ξεπεράσουν τους χρόνους οδήγησης, πράγμα που ε, απειλεί την ασφάλεια και γι' αυτό πολλές φορές τηλεφωνάνε με τα κινητά τους και ζητάνε παρακαλώ ελέγξτε μας μόλις τώρα που θα φτάσουμε εκεί αλλά θα πρέπει όμως να μην κοστίζει ο έλεγχος τόσο πολύ χρόνο. Το θέμα της επικροτικότητας και της κρατικής ενίσχυσης ε, ε, παίζει βέβαια ένα ρόλο. Το θέμα της ε, υποδομής των ε, θέσεων για πάρκινγκ, αυτό είναι θέμα υποδομής του κράτους μέλους. Εμείς θα το πληρώσουμε όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πού χρησιμοποιούν τα χρήματα, πού γίνονται οι επενδύσεις. Καταρχήν λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα με την έκθεση αυτή, εκτός από τις λίγες παρατηρήσεις που σας παρουσίασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ ως εισηγητής της ε, ομάδας μου θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της που μέχρι στιγμής ε, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι μπόρεσε να συνενώσει όλα αυτά τα πολλά στοιχεία. Και κατά βάση έχουμε εδώ τώρα τους ε, λόγους για τους οποίους δεν λειτουργεί το σύστημα όσο θα έπρεπε. Ακριβώς λόγω των πολύ ασαφών διατυπώσεων του μέχρι του δεκανονισμού και ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη να έχουμε μια νομική δέσμευση. Σε γενικέ γραμμέ ε, στηρίζω την άποψη τη εισηγήτρια. Θα ήθελα να μην αναφερθώ σε κάθε συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε τρία συγκεκριμένα σημαντικά. Καταρχήν, τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στο, όσον αφορά το είδος και το ύψος των κυρώσεων που πρέπει να μειωθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ύψος των προστήμων του υψηλότερου και του χαμηλότερου θα πρέπει επίση να καθοριστεί και όπως και η συνάδελφος Ράνερ, έτσι και εγώ θεωρώ ότι με το άρθρο 83 παραγραφος 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε ένα μέσο για να μπορέσουμε στο μέλλον να κινηθούμε προς σωστή κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου, αυτό που θα πρέπει ακόμα να συζητηθεί είναι η δημιουργία αυτής της λεγόμενης υπηρεσίας. Η στόχοι που ανέφερε η συνάδελφος Ράνερ είναι σωστοί νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον αυτή η υπηρεσία χρειάζεται πράγματι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε και τι γίνεται με το θέμα της εκπαίδευσης των λεγόμενων ελεγκτών, το να υπάρχουν πιο συχνή έλεγχοι και πιο εις βάθος κλπ. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει και ένα φυλάδιο σε όλες τις γλώσσες της ε, Ένωσης ενημερωτικό Από την άλλη μεριά εγώ θα έλεγα ότι τα μέσα που υπάρχουν με στιγμή που έχουν συστατικό χαρακτήρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και τις μεθόδους που υπάρχουν 2003-45 παραδείγματο χάρη ένα κανονισμό που μας δίνει τη δυνατότητα να ε, έχουμε κάποια κατευθυντήρια γραμμή. Οπωσδήποτε το σημαντικό είναι να είναι δεσμευτικά νομικά όλα αυτά τα μέτρα και είμαι σίγουρο ότι στο μέλλον θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ την συγκήτρια. Είχα όμως μία απορία και ένα σχόλιο. Η απορία. Δεν είναι δύσκολο να επεξεργαστεί κανείς αυτό το ψήφισμα από τη στιγμή που υπάρχει η οδηγία, η προηγούμενη οδηγία που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη και η συνθήκη της Λισαβόνας που αλλάζει τα πράγματα και δίνει μεγαλύτερα περιθώρια διευθετήσεων ενώ παράλληλα υπάρχει και κάποια σύγχυση για τα εθνικά, για τις εθνικές υπηρεσίες καθορισμού των διαδρομών. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα ακόμη ασαφή και ασταθή. Και αυτό κάνει τα πάντα δύσκολα. Και το σχόλιο είναι ότι Μπορεί κάποια έκθεση να γίνει πρόφαση για άλλες. Σε αυτή τη συγκεκριμένη, αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία ή η μεγαλη υπηρεσία υπήρξε προηγουμένως για τις οδικές μεταφορές και είδαμε ότι το πρόβλημα είναι τι συνέχεια δίνεται, τι δίωξη υπάρχει για τις διαμεθοριακές παραβιάσεις. Η υπηρεσία και οι διώξει λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα συνδυάζονται. Αυτό φάνηκε και σε άλλες περιπτώσεις και κάποτε θα χρειαστεί μάλλον να τα δούμε και αυτά. Να το ξανασκεφτούμε τουλάχιστον πέρα και από αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα όρια του θέματος. Στούμε Σαλέτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ήρθα από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμών, όπου ψηφίσαμε 370 τροπολογίες για τον έλεγχο του προπολογισμού 20 διαφορετικών ευρωπαϊκών οργανισμών. Και πρέπει να πω ότι όταν ακούω να μιλάμε για τη δημιουργία μια επιπλέον υπηρεσίας, ενός επιπλέον οργανισμού, τρομάζω. Σκέφτομαι τους ε, Ευρωπαίους φορολογούμενους και το εκλογικό μα αιώμα, το οποίο φυσικά δεν θα ακούσει με ικανοποίηση τη δημιουργία ενό ακόμα ευρωπαϊκού οργανισμού. Και αυτό φυσικά θα τροφοδητήσει και επιπλέον ευρωσκεπτικισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράνε, η οποία ετοίμασε ένα πάρα πολύ καλό κείμενο και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να πω και συμφωνώ και με τους δύο προλαλήσαντες που αναφέρθηκαν στο Γκαλιλαίο και στο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης. Ε, όλα όσα έλεγε ο συνάδελφος είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αν και εγώ ε, ως εκπρόσωπος ε, μιας χώρας που ε, προσφάτως προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να μιλήσω και για τις αρχές εφαρμογής. Η χώρα μου είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το 2008 συνεισέφερε στο σύστημα αυτό ε, και η συνεισφορά ήταν μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε και πραγματικά αυτό μου φαίνεται παράδοξο και πρέπει κάτι να γίνει από αυτού. Ευχαριστώ κύριος Πασκουαρέλη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν δέχεται την έκθεση αυτή και θα μπορούσαμε να πούμε ότι γενικά υποστηρίζουμε όλες τις ιδέες που εκφράζει δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφωνία εκτός ίσως από την υπηρεσία. Μέχρι προσφάτως υπήρχε σαφής περιορισμός στο τι μπορεί να κάνει η Ένωση, στο τι μπορούσε να κάνει η Ένωση για την επιβολή της εφαρμογής των ίδιων της των κανόνων. Δεν υπήρχε δηλαδή καμιά δικαιοδοσία για εναρμόνιση κυρώσεων ή διώξεων, τουλάχιστον για τις μεταφορές, τις υδροδρομικές. Από τότε όμως έχουν γίνει πολλά από την Κομισιόν ώστε να υπάρξει μια κοινή ερμηνεία των κανόνων. Αυτό σε συνεργασία με εθνικές επιτροπές με τις οποίες συζητήσαμε πολλά για λεπτά και δύσκολα προβλήματα του κανονισμού οι σημειώσεις αυτές θα έχουν δημοσιευτεί και στο ίντερνετ και αλλού, είναι γνωστές ως κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ελήφθηκε μια απόφαση για την τυποποίηση ή ταξινόμηση των κυρώσεων. Προσπαθούμε δηλαδή με τα κράτη-μέλη, μαζί με τα κράτη-μέλη να δούμε ποιες παραβιάσεις είναι οι σοβαρότερες και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Και ποιες άλλες μπορούν να θεωρηθούν ως πλημελήματα. Επίσης, η συνθήκη της Λισαβόνας πράγματι ανοίγει καινούριου δρόμους για εναρμόνιση του ποινικού δικαίου το άρθρο 83 όπως υπόθηκε αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει η Κομισιόν να κάνει καταρχάς πρόταση και αντί να τροποποιεί κανόνες που έχουν εγκριθεί μόνο 3-4 χρόνια πριν για μας προτεραιότητα είναι η σωστότερη εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων. Αυτό το κάνουμε μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που καθίσταται δυνατή και από τους κοινωνικούς κανόνες την αρχή δηλαδή την αρχή της ετεροδικίας όπου βάσει της οποίας μπορεί μια χώρα να επιβάλλει κυρώσεις και για δίκημα που διεπράχθη σε άλλη χώρα μέλος μέσω του ψηφιακού ταχογράφου παραδείγματος χάρη και πρόσφατα η λεγόμενη οδική δέσμη καθόρισε εθνικά μητρώα αρχεία για τις παραβιάσεις που σημειώνονται από οδικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οδικών μεταφορών. Όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο της ε, πολιτικής μεταφορών, οδικών μεταφορών, που στοχεύει στη διπλή ασφάλεια και των προσώπων και των αγαθών. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα πειραματικά ή πιλωτικά προγράμματα με τα οποία ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι όταν θα δημιουργούν νέες υποδομές, θα διαχειρίζονται τις παλιές, θα διασφαλίζουν επίσης ότι όλα αυτά γίνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια εκείνων που πρέπει να εργάζονται όπως τους οδηγούς, να υπάρχουν τόποι αναπαύσεως για να γίνεται σεβαστή και η κοινοτική νομοθεσία. Τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν τώρα για αυτό το πρακτορείο ή την υπηρεσία οδικών μεταφορών η Κομισιόν όπως ξέρετε έχει αποφασίσει για τις ζώνες ασφαλείας να γίνουν αυστηρότεροι κανόνες και υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών οργάνων για το ρόλο των υπηρεσιών αυτών μέσα στην Ευρώπη γενικότερα γιατί δεν έχουμε κάνει καμία πρόταση για νέες υπηρεσίες, όχι γιατί πρόκειται για χάος, όπως ήθελε να πει ο κ. Μπράντορν, πράγμα το οποίο μπορεί να ισχύει για τη χώρα του, αλλά γιατί οι υπηρεσίες που έχουμε εμείς στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών είναι πολύ επαγγελματικές και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτές. Τέλος, η κυρία Χάνα λέει ότι θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει και αυτό ένα ρόλο αν αποφασίσει η Κομισιόν ότι πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός των ελέγχων. Ξέρετε ότι όπως έχει νομοθεσία προβλέπει ότι η έλεγχη επιτόπου στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αλλά και στους δρόμους πρέπει να δείχνει μάλλον, δείχνει ότι αυξάνονται και μάλιστα καμιά φορά και κατά 4% οι, αριθ, οι μέρες οδήγησης των οδηγών και αυτό είναι πολύ μεγάλος αριθμός και όταν θα ξεπεραστεί το το φορτηγό που θα διαθέτουν τον ε, ψηφιακό ταχογράφο. Θα τα δούμε όλα αυτά λεπτομερέστερα. Θα δούμε καταρχήν αν έχουμε φτάσει το 90% και αν ναι τότε θα μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις από το 3% να περάσουμε στο 4% των ελέγχων. Και αυτό φυσικά θα υποβληθεί και στο Κοινοβούλιο μέσω της κανονικής συνήθως διαδικασίας επιτροπολογίας. Φυσικά θα πληροφορηθεί εν καιρό στο Κοινοβούλιο, εν καιρό το δέοντι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υποθυμίσω ότι δεν υπάρχει πια επιτροπολογία ως όρος. Ναι, ναι. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ για τις σημαντικές συμβολές. Νομίζω ότι ε, όσον αφορά τους στόχους που επιδιώκουμε δεν διαφωνούμε καθόλου. Θέλουμε ασφάλεια στους δρόμους, θέλουμε την προστασία των εργαζομένων και λειτουργών συστήμα στις δικές μεταφορές. Είναι αδύνατο εδώ να πούμε ότι μια μέρα στην άλλη, στην ό,τι θέλουμε. Σε όλα τα τη μια υποδομή που προσφέρει την ίδια ασφάλεια. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να το πετύχουμε βήμα προς βήμα. Υπάρχουν σε ορισμένε χώρε ε, απαρκώς ε, ικανοποιητική υποδομή, σε άλλες όμως υποδομή που θα πρέπει να βελτιωθεί. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Εγώ δεν είμαι τώρα υπέρ μιας νέας υπηρεσίας, δηλαδή να λέμε άμα δεν φανταστούμε τίποτα καλύτερο, δημιουργούμε μια υπηρεσία και λύνουμε τα προβλήματά μα. αλλά μετά από πολλέ συζητήσει είδα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του αλλιώ στην πράξη δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσαρμογής των συστημάτων. Θέλω πρέπει να ξέρω τι γίνεται σε άλλε χώρε, γιατί ορισμένε χώρε έχουν πολύ καλέ μελέτε, πολύ καλά στοιχεία, άλλε, όχι τόσο. Και τώρα, κατά πόσο θα πρόκειται για μια υπηρεσία ε, που θα είναι ανεξάρτητη, θα ε, εναχθούμε σε κάποια άλλη ισχύουσα και υπάρχουσα η υπηρεσία. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε ένα βήμα επικοινωνίας και ανταλλαγή πληροφοριών. Εγώ θέλω οι καθημερινές γραμμές που υπάρχουν ήδη να αποστούν δεσμευτικές και να είναι κατανοητές για όλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Και ένα τελευταίο πρόβλημα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. πολλοί που κυκλοφορούν στους δρόμους μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προέρχονται από τρίτες χώρες. Δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία που και τα συστήματα που λειτουργούν σε εμά. Ε, κατάλληλη πληροφορία λοιπόν που θα ενημερώνει τους οδηγούς αυτούς ε, τι σημαίνει το ότι μπαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρω αυτό από οδηγούς που έρχονται από ανατολικέ χώρες και περνάνε από όλη την Ευρώπη και δεν μπορούμε να προϋποθέτουμε ότι γνωρίζουν τους κανόνες μας και θα πρέπει γι' αυτό με ε, ε, κατανοητό τρόπο να τους παρουσιάσουμε τις διατάξεις που θα πρέπει να τηρούν όσων κινούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το, καταφέρουμε αυτό με αυτό το, το φάκελο που έχουμε μπροστά μας, θα είναι πάρα πολύ καλό και θα έχουμε αυξήσει την ασφάλεια στους δρόμους εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Θα χαρώ να έχω πολλές καλές τροπολογίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γλίγορα με την νομοθεσία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ράνε. Να ενημερώσω τα μέλη για την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 6 Απριλίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή τις 27 και 28 Απριλίου και προβλέπεται να πάμε στην Ολομέλεια το Μάιο. Προθεσμία τροπολογιών 6 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσε η πρωινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Συνεχίζουμε στις 3 ακριβώς με τον Ισπανό Υπουργό. Ευχαριστώ.